Dear colleagues, open Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίασή μας. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκρισή της. Υπάρχουν παρατηρήσεις παρακαλώ. Δεν βλέπω παρατηρήσεις. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Και έχω πολλέ. Προσέξτε με λοιπόν. Πρώτον, συστάσεις και αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνάντηση των συντονιστών 11 Πέμπτου ότι η σημερινή μας συνεδρίαση παρατείνεται κατά 30 λεπτά. Αν και αναβλήθηκε η εκθέση Μπέρες, ορισμός μελών, IFRS, πρέπει να αποφασιστεί συγητής αργότερα. Αποφασίστηκε ότι στις 25 Ιουνίου πρέπει να πάει στο ΑΕΣ στη Ρήγα. Ορισμοί επίσης εκθέσεις την οδηγία την έχουν πάρει πράσινη ανταλλαγή απόψεων επίσης για φορολογία. ...2348 οδηγία για την φορολογία... Ε, το S&D πήρε για τη, τα επιτόκια και έκθεση για την Τραπεζική Ένωση ή Σοσιαλιστές 2014 της έκθεση για τον ανταγωνισμό του ΕΛΚΑ και γνωμοδοτήσεις προπολογισμός 2016 όλα τα τμήματα κανείς δεν ήθελε το θέμα αυτό οπότε ο Ρομπέρτο θα το αναλάβει πολύ θα χαρεί 2014 η επιετήσια έκθεση η ΓΚΟΕ. Οικονομική διακυβέρνηση. Οι συντονιστέ είπαν ότι θα έχουμε μεικτή συνεδρίαση στη... τον Ιούνιο με την ε, απασχόληση για να έχουμε οικονομικό διάλογο με τον Αντιπρόεδρο Τομπρόφσκι, την κυρία Τάισεν και τον κύριο Μοσκοβισή για τι συστάσει στι ειδικέ αναχώρε. Επειδή δεν υπάρχει ο χρόνο, οι συντονιστέ αποφάσισαν να μην συντάξουμε γνωμοδότηση για την έκθεση για γραμμές γραμμέ για την απασχόληση τη Επιτροπή Απασχόληση. Σα στείλουμε επιστολή στον κύριο Σούλ ζητώντα συζήτηση στην Ολομέλεια να γίνει στα πλαίσια τη ε, κρίση και να έχουμε και εκπροσώπου από την ελληνική κυβέρνηση. Όσον αφορά το ΕΦΣΥ. Τριμερίος διάλογος έλαβε χώρα τον προηγούμενο μήνα, τελείωσε στις 3 το πρωί. Ελπίζω να είχαν καλό καφέ. Όλα τα θέματα τώρα έχουν καλυφθεί και έχει επιτευχθεί πρόοδος. Άλλα σημαντικά θέματα πρέπει να αποφασιστούν ακόμα με το Συμβούλιο, ιδιαίτερα τη έκπληξη για τη χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ και για την διακυβέρνηση, για το επενδυτικό ταμείο του Juncker δηλαδή. Θα γίνουν και δύο επόμενοι τριμερείς διάλογοι σήμερα, γι' αυτό και ο Ρομπέρτο δεν είναι εδώ, ούτε και κάποιοι συνάδελφοι. Και προβλέπεται και ένας ακόμα για αύριο το βράδυ. Και ελπίζω να έχουν καλύτερο καφέ από ό,τι έχουμε στο Στρασβούργο, λέει ο πρόεδρο. Για τι κεφαλαρακορκιδές. 26 Φεβρουαρίου αποφασίστηκε ο φάκελο αυτός να πάει στην Ολομέλεια πριν τι τριμερεί διαπραγματεύσεις. 29 Απριλίου ψηφίσαμε, ε, άλλη επιτροπή, η ΚΟΝ θα ψηφίσει βάσει εντολή τη Ολομέλειας. Ω ήθιστε, οι διαπραγματευτές είναι ο συγητής, οι σκιώδης και θα αρχίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα εφόσον το Συμβούλιο έχει εγκρίνει τη δικιά του γενική προσέγγιση. Ως ήθιστε, περιμένουμε το Συμβούλιο. Για τα benchmark, η ΕΚΟΝ έκανε την έκθεσή της στις 31 Μαρτίου και αποφάσισε να πάει στην Ολομέλεια ο φάκελος για ενισχυμένη εντολή για διαπραγματεύσεις με τριμερή διάλογο. Η Ολομέλεια ψήφισε στις 19 Μαΐου και αποφάσισε να επανεπευθεί στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 61 του κανονισμού. Οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Επιτροπή λοιπόν μπορούν να αρχίσουν πλέον βάσει εντολή τη Ολομέλεια. Ω ήθιστε, η διαπραγματευτική ομάδα έχει ήδη καθοριστεί. Ο πρώτο τριμερή διάλογο προβλέπεται για τι 2 Ιουνίου. Αυτά περί benchmark. Το Συμβούλιο είναι έτοιμο δηλαδή. Και το τελευταίο, δεύτερο τριμερή διάλογο για την ασφάλεια των οικονομικών συναλλαγών ο δεύτερο τριμερή διάλογο για το σχέδιο κανονισμού αυτού έλαβε χώρα στι 20 Μαου και μπορώ να σα πω ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδο, οπότε τα περισσότερα θέματα θα μπορέσουν να συζητηθούν στον τριμερή διάλογο και να καταλήξουν. στι 3 Ιουνίου δηλαδή. Όσον αφορά τι εξαιρέσει για τι κεντρικέ τράπεζε, έχει επιφυλάξει στο Συμβούλιο για την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ροή δεδομένων και πρέπει να υπάρξει τεχνική δουλειά όσον αφορά τις δυνατότητες Επιτροπής να επεκτείνει τις εξαιρέσεις στις κεντρικές τράπεζες των χωρών. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις αναφορές, το Συμβούλιο εκφράζει ανησυχία για τις προτάσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις Backloader και τα θέματα αναφοράς. Για τις εξαιρέσεις όσον αφορά την υποχρέωση αναφοράς και το phase-in, οι διαπραγματευτές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσει το 117 και 118 και να πάει σε τεχνικό επίπεδο η συζήτηση. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφάσισαν ότι το τεχνικό επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιήσει το άρθρο 15, αλλά επιμένει στο δικαίωμα των χωρών μελών να προχωρήσουν σε πιο φιλόδοξες διατάξεις. Ο επόμενο πολιτικό τριμερή διάλογο θα καλύψει παρετέρω θέματα όπως είναι η διαφάνεια, οι εκθέσεις των επενδυτών, οι υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού και επειδή δεν υπήρξε επαρκής πρόοδος στον προηγούμενο τριμερή διάλογο, ούτε στις χώρες, έχει συνεχιστεί η τεχνική εργασία. Αυτά ήταν οι γενικές ανακοινώσεις. Παρατηρήσεις, παρακαλώ. Δημόσια κρόση τώρα σχετικά με τις συντάξεις. Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιδοτικών παροχών. We have uh, Έχουμε προσκαλέσει εδώ τον κύριο Σικάντσα από την Chance Europe. Πού είναι? Ναι, εδώ. Καλώς ήρθατε. Τον Hans Μέρτεν από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Τον Στίβμαν που είναι επικεφαλής της Aftergemeinschaft Γερμανία. Δεν καταλαβαίνω γερμανικά λέει ο πρόεδρος. Εντάξει. Λέει και ο κύριος Τσερούτη από την Business Europe. Ήρθατε όλοι, γιατί κάποιος μου είπε ότι κάποιος είχε μποτιλιαριστεί και δεν μπορούσε να φτάσει έγκαιρα. Προβλέπουμε μισή ώρα για τις παρουσιάσεις, για τους τέσσερις προσκεκλημένους μας δηλαδή, και μετά θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής μας. Πριν δώσω το λόγο λοιπόν στους ομιλητές μας, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για τις δραστηριότητε και την εποπτεία. Την πρόταση δηλαδή που έχουμε για την, ε, την κάλυψη ανακροπρόθεσμων ε, αναγκών χρηματοδότηση ευρωπαϊκής οικονομίας και πιο συγκεκριμένα τα στρατιωτικά ταμεία. Ο κύριος Χάγες. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια καλή συζήτηση. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Όπως ξέρετε, πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε μια πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή μας και ετοιμάσαμε και ένα μικρό έγγραφο. Σήμερα θέλουμε να ακούσουμε τον κλάδο, τους εμπειρογνώμονες, αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα όλον αυτό τον κλάδο. Δεν πρόκειται για συζήτηση στρογγυλή τραπέζης μεταξύ ρυθμιστών. Όχι. Θέλουμε να δούμε η πρόταση αυτή πώς θα επηρεάσει τα συνταξιδωτικά ταμεία, πώς θα επηρεάσει τον κλάδο στην Ευρώπη. Γι' αυτό θέλω πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να ακούσω τη σημερινή συζήτηση. Και επ' ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις. Θέλω να τους ακούσω, να ακούσω τις παρατηρήσεις τους όσο προχωρώ στην εκπόνηση της εκθεσής μου που θα είναι έτοιμη πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές μη σπαταλήσω περισσότερο το χρόνο μας. Θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, αν συμφωνείτε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε, Μπράιαν. Ο Τζον Σεγκάς, Pensions Europe. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα. Ε, με ιδιαίτερη ικανοποίηση συμμετέχουμε στην ακρόαση αυτή. Είναι καλό ο κλάδος, οι ευρωβουλευτές να συζητούν όσο γίνεται νωρίτερα στη διαδικασία. Ε, θέλουμε να βοηθήσουμε τον εισηγητή, τον κύριο Χάγια, τους σκιώδεις εισηγητές και τους άλλους ευρωβουλευτές για να υπάρχει πολύ καλός ο έλεγχος της πρότασης αυτής για την αναθεώρηση των κανόνων για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ταξιδότησης. Συμφωνούμε με τα όσα περιλαμβάνει το έγγραφο μελέτης που εκπονήσατε πρόσφατα και με τη στάση του εισηγητή. Στηρίζουμε επίσης και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έφτασαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να έχουμε ένα σταθερό, κατάλληλο και ασφαλές σύστημα συνταξιοδοτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος έχει αλλάξει μετά την πρώτη μορφή της οδηγίας που ήταν το 2003. Τα ταμεία μη επαγγελματική έχουν μεγαλώσει και έχουμε περάσει από το defined benefit στο defined contribution, δηλαδή από τις εγκυμένες συντάξεις στις συντάξεις για τις οποίες παίρνει μέρος του κινδύνου και ο ίδιος ο δικαιούχος. Η νομοθεσία συνεπώς, πρέπει και αυτή να αλλάξει. Μας ικανοποιούν οι προτάσει που βλέπουμε όσον αφορά τη Solvency 2, τη χαρικιότητα 2, ότι ορισμένες κακές διατάξεις εκεί φεύγουν από τη μέση. Στόχος μας είναι η ασφάλεια, η καταλληλότητα, η διασημότητα των συνταξιδοτικών προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως είναι υπερβολικά λεπτομερές το Συμβούλιο προτείνει κάποιε απλοποίησει με περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή σε συνδυασμό με τα σταξιδωτικά συστήματα των χωρών μελών. Θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει το ίδιο. Με την ομάδα των 9, των ε, οργανώσεων δηλαδή, μεταξύ άλλων και της Business Europe και του ETGC, στείλαμε επιστολή στον εισηγητή και στους χιώδες εισηγητές όπου εξηγούμε την κοινωνική διάσταση των Ιδρυμάτων αυτών και γιατί χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. ρίνω λοιπόν την ε, Επιτροπή σας να το αναγνωρίσει αυτό σαν βασικό στοιχείο. Με τους κοινωνικούς εταίρους συνεργαζόμαστε και ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για κατανολωτικά προϊόντα. Και είναι σημαντικό επίσης να θυμόμαστε, όπως λέει και το έγγραφο εργασία σας, ότι οι συντάξει είναι εθνική αρμοδιότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το σημερινό πλαίσιο βέβαια είναι δύσκολο για τα συνταξιδοτικά ταμεία με χαμηλά επιτόκια, με πολλά αριθμιστικά επίπεδα. Υπάρχει επιπλέον πίεση λοιπόν στα συνταξιδοτικά ταμεία. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από τα ταμεία αυτά να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ρευστότητα μέσω των αγορών κεφαλαίων. Να επενδύουν ας πούμε σε ευρωπαϊκές υποδομές να δημιουργηθούν περισσότερε θέσει απασχόληση και να έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρούμε τη σωστή ρυθμιστική ισορροπία. Η ρύθμιση δηλαδή να μην ε, καταπολεμάει κάποιε από τι προσπάθειε που κάνουμε. Κάποια πεδία κλειδί λοιπόν τα οποία μπορούν να βελτιωθούν. Πρώτον, όσον αφορά το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Οι νέε απαιτήσει για τα επαγγελματικό προσόντα και για όλους ε, όσοι συμμετέχουν μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πια ονομαστικά τραστής και υπονομεύεται έτσι η κοινωνική συμμετοχή στα επενδυτικά αυτά προγράμματα. Δεν λέμε ότι δεν θέλουμε υψηλές προδιαγραφές ε, διακυβέρνησης, αλλά θέλουμε συλλογικά να γίνεται η αξιολόγηση και όχι μεμονωμένα. Πιστεύουμε ότι έτσι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Δεύτερον, η δήλωση ε, κερδών. Θα είναι πιο δύσκολο να δίνουν τα επενδυτικά ταμεία τις πληροφορίες που χρειάζονται. Θα γίνει πιο δύσκολη η δουλειά τους. Έχουν κάνει πολλές καινοτομίες τα τελευταία χρόνια τα επενδυτικά αυτά ιδρύματα. Χρησιμοποιούν τα οικονομικά στοιχεία έτσι ώστε οι δηλώσεις αυτές κερδών να είναι σαφείς για όλους. Αλλά έτσι όπως προβλέπετε τώρα θα ήταν αδύνατον οι ανακοινώσεις που θα γίνονται να εξυπηρετούν τα μέλη τους. Θα είναι σε βάρος ορισμένων μελών τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν περισσότερους κινδύνους σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Έπειτα τα διασυνοριακά ε, συνταξιδοτικά προγράμματα. Και εδώ υπάρχουν περισσότερες απαιτήσει. ή ενιαία η θετική αυτή μεταρρύθμιση μπορεί να είναι χρήσιμη εφόσον οι απαιτήσει χρηματοδοτούνται κατάλληλα. Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο. Για τις κατεξοδότηση πράξεις, κάποια τεχνικά ζητήματα στην οδηγία είναι ιδιαίτερα πολιτικά και πρέπει να αποφασίζονται δημοκρατικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει λόγο στον έλεγχο και όσον αφορά το DC deposit, δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τις επενδύσεις που προστατεύονται σε κάποιο άλλο σημείο της επενδυτικής αλυσίδας. Αλλιώς θα κοστίσει περισσότερα χρήματα που το κόστος αυτό θα πρέπει να το αναλάβουν τα μέλη, το οποίο έτσι καλώς θα πάρουν μικρές συντάξεις όταν ταξιδοτηθούν. Συνεπώς, προσοχή για το κόστος που επιφέρει η αναθεώρηση αυτή της οδηγίας. η έκθεση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται μόνο στο κόστος εφαρμογής της οδηγίας. Και λέει ότι είναι μόνο 27 αναμέλος ε, τον πρώτο χρόνο. Άρα τα μέλη θα πρέπει να τα πληρώσουν αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν το κόστος. Συνεπώς, στηρίζουμε την οδηγία, αλλά πιστεύουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί παρετέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Χάνς Φαν Μέρτεν έχει τώρα από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Thank Also... Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Καταρχήν να τονίσω κάποια αρχικά άρθρα των συνθήκων και το τι λένε για τις συντάξεις, καθώς και το πώς τις αντιμετωπίζει το ΔΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αυτές τις βασικές αρχές και τέλος θα τονίσω κάποιες ιδέες που μπορεί να ε, αποδειπούν χρήσιμες. Να ξεκινήσω με την ε, ε, απόφαση Φανχέντεν το 1962. Η ευρωπαϊκή κοινότητα δηλώνεται εκεί δημιουργεί ένα, μια νέα νομοθετική τάξη για την οποία οι τα ευρωπαϊκά κράτη ε, δίνουν την κυριαρχία τους για ορισμένα περιορισμένα ζητήματα ε, και δεσμεύουν ε, τα έθνη. Επίση, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι κανόνες περί ανταγωνισμού ισχύουν και για τα συνταξιδικά ταμεία στην, απόφαση στην υπόθεση Αλμπανή δηλώθηκε ότι το συνταξιδικό ταμείο που έχει αναλάβει την τροποποίηση ενός ε, επικουρικού ταμείου γίνεται αυτό μέσα στη, σύμφωνα μάλλον με το νόημα της συνθήκης. Επιπλέον το 2011 άλλη απόφαση ε, δηλώνει ότι η ελεύθερη προσφορά υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών ισχύει για τα συνταξιδικά ταμεία και αυτό σε σχέση με τις επαγγελματικές συντάξεις πρόκειται για υπηρεσίες με την έννοια του άρθρου 75 της συνθήκης. Υπάρχουν προβλέψεις όσον αφορά τις άμοιβες, ε, τις αποζημιώσεις και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζονται αυτού του είδους οι υπηρεσίες. Την ίδια απόφαση επίσης λέγεται στο σημείο 38 ότι επίση θα πρέπει να δηλώσουμε ότι από την οπτική της ενιαία αγοράς και έτσι ώστε να επιτεθούν οι στόχοι αυτής της ενιαία αγοράς, το άρθρο 65 ε, της ε, οδηγίας περιπηρεσιών αποκλεί οποιοδήποτε εθνική ε, ρύθμιση που μπορεί να επηρεάσει και να επιδεινώσει την παροχή υπηρεσίας εντός κράτους ή ανάμεσα σε δύο κράτη. Αυτά είπε το δικαστήριο, το 10. Επίσης το 2011 το δικαστήριο μίλησε για κρατική ευθύνη για την μη τα μη λειτουργούντα συνταξιδοτικό ταμεία ε, στην υπόθεση Όλμπαρτ ε, αποφάσισε ότι η οδηγία 2008 του 89, δηλαδή αφαιρεγγιότητα, δεν έχουν επιφέρει το αποτέλεσμα που, θέλουν, που ήθελαν οι καταγγέλλοντες. και οδήγησε σε μείωση των δικαιωμάτων τους, δηλαδή παράβαση των υποχρεώσεων του κράτους μέλους. Με άλλα λόγια, η κρατική ευθύνη, η εθνική ευθύνη, αν φτάσουμε το επίπεδο το 49% ισχύει ε, και τότε το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο επειδή δεν έχει επιδειχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν για, τους για τα μη λειτουργώντα ε, ε, ε ταμεία ευθύνεται το κράτος. Και θα ήθελα να μεταβώ τώρα στο θέμα της ε, Ένωσης ε, των Κεφαλαιογορών και τη σχετική πρόταση. Εγώ την εξέτασα και ε, εκεί τονίζεται 18 φορές η λέξη συντάξει, συνταξιωτικά ταμεία. Δηλώνεται ότι η άρση των εμποδίων στη, για τη διασυνοριακή αγορά μπορεί να ε, περιορίσει τις, τε, τις σχέσεις των συνταξιωτικών ταμείων. Και δεν ξέρω ποια θα είναι η σχέση ανάμεσα σε αυτό και την ε, ε, οδηγία περί συνταξιωτικών ταμείων 2. Επίσης είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ότι στην Solvency 2, στην Αυτοκυριακότητα 2, έχει, υπάρχει το άρθρο 204 το οποίο λέει ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ένας όμιλος και το συνταξιδικό ταμείο είναι ένας όμιλος, μια επιχείρηση, ε, ισχύουν μόνο στο κράτος όπου έχει εγκριθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ε, Άρα λοιπόν μπορούμε να αποκομίσουμε τέσσερα διδάγματα από από όλα αυτά. Καταρχήν πιστεύω ότι η εναρμόνιση των κεφαλαγορών είναι απαραίτητη ώστε να παρεμποδιστεί η ρυθμιστική διαιτησία, αρμπιτράζ. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, είτε η ΑΙΟΠΑ θα ενεργεί μόνη τη, όπως το βλέπουμε τώρα, πράγμα που με τη σειρά του θα αρχίσει να ισχύει ούτως ή άλλως, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι για τις διασυνοριακές δραστηριότητες των συνταξιδικών ταμείων οι απαιτήσει κεφαλαϊκές είναι πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την αντιμετώπιση των κρατών μελών. Αν δηλαδή οι απαιτήσει διαφέρουν από κράτος σε κράτος, βλέπουμε ακριβώς την διατησία που θέλουμε εμείς να εμποδίσουμε. Δεύτερο δίδαγμα είναι ότι η οδηγία η θα πρέπει να καταστήσει ευχερέστερη και όχι δυσχερέστερη τη διασυνοριακή ε, παροχή υπηρεσιών. η διάταξη fully funded ε, είναι αυτή η οποία δυσχεραίνει περισσότερο τη διασυνοριακή λειτουργία των συνταξιδοτικών ταμείων. Ε, ο λόγος για τον οποίο ανέφερα το άρθρο Insolvency 2 είναι γιατί θα πρέπει να δούμε, να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις τοπικά δραστήριες εταιρείε και τις μη τοπικά δραστήριες. Ίσως αυτό να είναι μια επίλυση για το πρόβλημα το οποίο διαπιστώνουμε να υπάρχει, ότι δηλαδή πολλά συνταξιδοτικά ταμεία λένε γιατί να έχουμε όλους αυτούς τους κανόνες, ενώ μπορούμε να λειτουργούμε πολύ πιο φυσιολογικά Ήδη στον ε, ορισμό θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά και στη ε, ταμεία τα οποία λειτουργούν μόνο εντός των εθνικών τους ορίων. Να δούμε δηλαδή πώς ακριβώς θα πρέπει να φτιάξουμε τον ορισμό. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Για να κλείσουμε με όλα αυτά τα στοιχεία μαζί βλέπω ήδη τα θεμέλια μιας ένωσης ε, των συνταξιδοτικών ταμείων γιατί έχουμε κρατική ευθύνη, πράγμα που έχει ομοιότητες με τη Δραπεζική Ένωση και την Ασφαλιστική Ένωση και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τέτοια καταστροφή όπως με την κατάρρευση την πρόσφατη των, της οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μέρτεν. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Κλάου Στίβενμεν που είναι... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη τιμή για την οργάνωσή μας, ABA, που μας προσκαλέσατε εδώ. Εμείς υποστηρίζουμε την διαδικασία της αναθεώρησης και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και εμείς να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η οδηγία IORP. Οι επαγγελματικές συντάξεις έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όταν συγκριθούν με ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αυτό έχει λεχθεί και πριν είναι χαμηλότερο το δυτικό κόστος, η κατανομή του κινδύνου και μέσα στην ίδια γενεά αλλά και μεταξύ γενεών βελτιώνει το, είναι βελτιωμένη και βελτιώνει και το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι περίπου 60% των Ευρωπαίων εργαζόμενων δεν καλύπτονται ακόμη από επικουρικές συντάξεις. Κάτι που στο μέλλον στις χώρες που θίγονται θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Χρειαζόμαστε καλύτερο μείγμα των προβλέψεων για τη ταξιοδότηση. Γι' αυτό χρειάζεται να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς με την οδηγία IORP 2 για τις επαγγελματικές συντάξεις και η IORP αυτή τη στιγμή είναι μέρος μόνο των επαγγελματικών συντάξεων και να τους επιτρέψουμε λοιπόν να λειτουργήσουν. Θέλω να τονίσω ακόμη ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούμε να έχουμε συστήματα τριών πυλώνων. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές φιλοσοφίες, νοοτροπίες, διαφορετικά ιστορικά υπόβαθα. Δεν υπάρχει αυτό που λένε στα αγγλικά one size fits all. Δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις πουθενά. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ο χώρος για ε, λύσεις για τις ευικουρικές συντάξεις του τύπου one size fits all. Η ενότητα βρίσκεται μέσα στην ποικιλομορφία και αυτό ισχύει βεβαίως και για τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι επαγγελματικές συντάξεις παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κοινωνική ασφάλεια. Βεβαίως είναι τα προγράμματα που τις παρέχουν είναι νομικές οντότητες, αλλά είναι σημαντικά σε ένα χώρο όπου εργοδότες και εργαζόμενοι και IOP εμπλέκονται. Πρόκειται για ένα τρίγωνο δηλαδή που αυτό επιφέρει την διαφορά. Δηλαδή δεν είναι απλά συνταξιοδοτικά ιδιωτικά προγράμματα. Ε, εξακολουθεί δηλαδή ο εργοδότης στη Γερμανία, στη γερμανική νομοθεσία, να ε, στηρίζει το σύστημα αυτό. Εμείς έχουμε στη Γερμανία προστασία για την αφαιρεγγιότητα, προβλέπεται δηλαδή, επομένως δεν καλείται ποτέ το δημόσιο να καλύψει ε, ελλείμματα των συστημάτων αυτών. Αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει και το blueprint για όλη την Ευρώπη. Από το 1974 ούτε μία περίπτωση δεν είχαμε στη Γερμανία όπου ένας απασχολούμενος ή δικαιούχος να μην έχει λάβει τα υπεσχημένα ακόμα και αν υπήρξε πτώχευση της εταιρείας που στήριζε το συνταξιδοτικό του πρόγραμμα. Όπως είπα, ε, είμαστε ενωμένοι στην ποικιλομορφία και γι' αυτό χρειαζόμαστε μοναχά ελάχιστα στάνταρτ. Δεν χρειαζόμαστε οποιαδήποτε εναρμόνιση των συστημάτων. Και δεν συμφωνώ ότι αυτό συμβαίνει, ε, ότι μάλλον λόγω IOP 1 δεν έχουμε τόσο πολλές διαμεθοριακές επιχειρήσεις για τα συνταξιδοτικά. Δεν χρειάζεται μάλλον, διότι τα συστήματα επικουρικών συντάξεων λύνουν εθνικά συνταξιδοτικά προβλήματα. Όσο δεν έχουμε ενοποιημένο ευρωπαϊκό πρώτο πυλώνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ενοποιηθεί ο δεύτερος ή ο τρίτος πυλώνας. Για το λόγο αυτό πιστεύω ακόμη ότι οι απαιτήσει της Solvency 1 που έχουμε έχουν αποδώσει, έχουν κάνει τη δουλειά τους. Αν θέλετε να βελτιώσετε τα πράγματα ακόμη περισσότερο, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ήδη αναφέρθηκαν ορισμένα από αυτά. Αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι οι επικουρικές συντάξεις πρέπει να υπακούν στα εθνικά κοινωνικά δίκαια και δίκαια εργασίας. Δεν είναι θεσμοί του τρίτου πυλώνα και γι' αυτό δεν υπάρχει χώρος για πράγματα όπως προστασία καταναλωτών γιατί στη Γερμανία όπου για παράδειγμα σύμφωνα με το δίκαιο ο εργοδότης υπόσχεται την επικουρική σύνταξη καταναλωτής είναι ο εργοδότης και όχι ο εργαζόμενος. Γι' αυτό και πρέπει νομίζω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλους τους τομείς που ενδέχεται να προκαλέσουν έξτρα δαπάνες και έξτρα επιβαρύνσεις. Ξαναλέω, 60% των Ευρωπαίων εργαζομένων δεν έχουν επικουρικές συντάξεις. Ακόμα και στη Γερμανία έχουμε 40% χωρίς και το 60% που έχει τέτοιου είδου σύνταξη στη Γερμανία δεν είναι αρκετά υψηλή η σύνταξη αυτή. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μην προκαλέσουμε περαιτέρω επιβαρύνσεις, αλλά να ανοίξουμε καλύτερα το δρόμο για να λειτουργήσουν τα συστήματα των επικονικών συντάξεων. Ο κύριος ε, Φέρμπερ, Προεδρεύον, ευχαριστώ κύριε Στίφερμαν και τέλος Μάξιμ Τσερούτη, ε, τη της Business Europe. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχετε στην ακρόαση. Ίσως όπως έγινε και με άλλα έγγραφα εργασία του εισηγητή σε αυτήν την Επιτροπή, πιστεύω πως είναι σημαντικό να θυμόμαστε ε, το, το θέμα το οποίο εξετάζουμε. Οι IOPS ε, αντιπροσωπεύουν 2,5 δις ε, ε, είναι το 25% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτά τα ταμεία, αλλά σίγουρα σε ορισμένα κράτη-μέλη πρόκειται για ήδη ανεπτυγμένη πρακτική. Οι εργοδότες παρέχουν επαγγελματικές συντάξεις και μετά σε επίπεδο της ευρωπαϊκό, η Business Europe είναι η φωνή των επιχειρηματιών και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Το σημαντικό κλειδί είναι για μας ότι αυτά τις επαγγελματικές συντάξεις θα πρέπει να παρέχονται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Όταν λοιπόν εξετάσουμε το πρόσφατο παρελθόν, η σημασία αυτών των ταμείων αυξάνεται. Είδαμε τις εξελίξεις ε, επιτόπου από τα επιδόματα στη, ε, στη συμμετοχή, δηλαδή στην ανάληψη μέρους του κινδύνου από τους δικαιούχους τους ίδιους. Πολύ σημαντική εξέλιξη και ελπίζουμε ότι στο μέλλον αυτό θα στηρίξει την ε, αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των ε, συνταξιωτικών ταμείων. Γι' αυτό εμείς ως Business Europe συμμετέχουμε με την στήριξη και των συνδικάτων, διότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα ε, ώστε να έχουμε ένα σωστό πλαίσιο και ε, τα επαγγελματικά, οι επαγγελματικέ συντάξει ως τμήμα όλων των αστεξιωτικών ε, πυλώνων και δομών θα παίζουν το ρόλο του πλήρω. και θα υπάρχει φυσικά δυναμικό για εξέλιξη, για ανάπτυξη σε όλε τι χώρε, ώστε να εξυπηρετηθούν αυτέ οι ανάγκε. Για να έχουμε όμως περισσότερους εργοδότες που θα παρέχουν επαγγελματικές συντάξεις με αποτελεσματικό τρόπο πρέπει να έχουμε στο κατάλληλο πλαίσιο έχουμε στόχους να σεβαστούμε τον κοινωνικό στόχο των επαγγελματικών συντάξεων και να εξασφαλίσουμε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση των συστημάτων πρόκειται έπειτα για μια συλλογική ε, πρωτοβουλία ως τμήμα της σχέσης ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο και δεν είναι ατομική ε, ενέργεια. Έπειτα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα εξουδεξιωτικά ταμεία θα παραμείνουν εθνική αρμοδιότητα, να αποφύγουμε την ε, την ενιαία προσέγγιση για όλους την UNICEF τρίτος στόχος είναι να αποφύγουμε νέα, νέους κανόνες όσον αφορά τις κεφαλαϊκές υποχρεώσεις γιατί αυτές ε, επιφέρουν κόστος, πράγμα που σημαίνει ε, δυσχέρεια για τους εργοδότες να παρέχουν τέτοιες επαγγελματικές συντάξεις και αυτά τα μέτρα δεν αιτιολογούνται μέσω της, από την ανάγκη να υπάρξει ισότιμο πεδίο ανάμεσα στα παραδοσιακά συνταξιδικά ταμεία και τα επαγγελματικές συντάξεις. Ε, γιατί παίζουν με διαφορετικούς τα, κανόνες ούτως ή άλλως, γιατί πλήρουν άλλο ρόλο, όπως είπαν και οι προηγούμενοι μιλητές. Εμείς στηρίζουμε το σχέδιο γνώμης της Επιτροπής Απασχόλησης του Κοινοβουλίου για να μην εφαρμόζονται πλήρως χρηματοδοτούμενες απαιτήσει στις διασυνοριακές παροχές τέτοιων συντάξεων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είναι υπερβολικά λεπτομερείς οι απαιτήσει γιατί πιστεύω ότι μια εναρμονισμένη δήλωση τέτοιων ε, συνταξιδοτικών επιδομάτων δεν αφήνει χώρο για τη συνέχιση των ε, διαφόρων θεμητών εθνικών ε, διατάξεων που υπάρχουν. Το Συμβούλιο ως προς αυτό έχει κάνει κάποια πρόοδο, αλλά χρειάζονται και περισσότερα βήματα. Βασικό μας μέλημα είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσει για τα συνταξιδικά ταμεία δεν θα είναι ομοιόμορφες, δεν θα, είναι, ε, δεν θα υπάρξει εκεί εναρμόνιση. Το είπαμε και παλιότερα ε, εδώ όταν ε, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την προστιθέμενη αξία των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η συζήτηση αυτή λοιπόν έχει ήδη γίνει σε διάφορες επιτροπές και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Απασχόλησης. Η θέση που ελήφθη τότε θα πρέπει να κυριαρχήσει κατά τη γνώμη μας, αλλά βλέπουμε ότι στο σχέδιο της Κομισιόν με το αναξιολόγηση κινδύνου για τις συντάξεις που είναι σχεδιασμένο με παρόμοιο τρόπο με το Solvency Risk και το σχετικό πρότυπο, μπορεί να κινδυνεύσει μαζί με την εργασία που γίνεται στην ΑΙΟΠΑ με την ε, μελέτη ε, ποσοτικού αντικτύπου Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτά τα δύο στοιχεία, εάν μάλλον αυτά τα δύο στοιχεία συνδυαστούν, το πεδίο ανάπτυξης ε, για το μέλλον, για τις κεφαλαϊκές υποχρεώσεις ανοίγει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να περάσει από αυτήν εδώ την Επιτροπή ένα μήνυμα σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατανοεί γιατί ένα ψηλότερο κόστος για τις επαγγελματικές συντάξεις θα ήταν αντίθετο με τον πολιτικό ρόλο της αύξησης της παροχής επαγγελματικών συντάξεων. Γίνεται συζήτηση ωστόσο και στην Επιτροπή ε, Απασχόλησης και γίνεται πρόοδος και πιστεύουμε ότι γινόμαστε κατανοητοί. Η Business Europe, που αφού να αντιπροσωπεύει τους, εργοδότες, συνεργάζεται στενά με την, ε, τον κλάδο των συνταξιδοτικών ταμείων, επαγγελματικών συντάξεων και ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε έτσι να βρούμε λύσεις για την διασυνοριακή παροχή συντάξεων αλλά και για να συμβάλλουμε στην διασημότητα και την καταλληλότητα των συντάξεων. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πολύ Ο Πρόεδρος βέβαια στα αγγλικά. Βεβαίω είναι πολύ σημαντικό το θέμα αλλά έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα στην ημερησία διάταξη. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκα να παρέμβω. Τώρα έρχεται η σειρά των σκιωδών και όσων άλλων ε, μελών έχουν ζητήσει το λόγο. Πολ Τάγκ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους που προσήλθαν για να διεξαχθεί η συζήτηση που μου φαίνεται πολύ χρήσιμη. Ορισμένα από τα σχόλια αυτά, τα οποία έχω ξανακούσει, αφήνουν κάπως απορριμμένο. Λένε ορισμένοι από τους ομιλητές μας εδώ, μας αρέσει, δηλαδή καλοδεχόμαστε την οδηγία, μετά όμως απαριθμούν τα πράγματα στα οποία δεν συμφωνούν. Γιατί τέλος πάντων ε, καλοδέχεστε την οδηγία, τουλάχιστον αυτή την ερώτηση απευθύνω στον πρώτο ομιλητή, διότι για την ώρα δεν έχω κατανοήσει καλά. Το τονίζω αυτό διότι αυτό που επιζητούμε εμείς Δηλαδή ο ευρωπαϊκός στόχος που προσπαθούμε να επιτύχουμε με την οδηγία ποια είναι η ευρωπαϊκή διάσταση γιατί εδώ τέλο πάντων Ευρωβουλή είναι και είναι πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή που εξετάζουμε. Ε, αναζητώ λοιπόν τον ευρωπαϊκό στόχο αλλά μέσα από τα σχόλιά σας είναι δύσκολο να τον βρω. Τώρα πιο συγκεκριμένα Μόνο ένας μίλησε για regulatory arbitrage, για διατησία δηλαδή. Εγώ, ρυθμιστική διατησία εγώ βλέπω, για παράδειγμα, κάποιος φεύγει από Ολλανδία, πάει στο Βέλγιο, υπάρχει εκεί ανάγκη για τέτοια διαιτησία. Η οδηγία ΕΟΠΗ νομίζετε ότι κάνει αρκετά για να αποφύγει Τώρα υπάρχουν και διαμεθοριακές IORP και ε, εθνικές. Είναι πολύ πιο διαφοροποιημένη η προσέγγιση. Και πρέπει να ε, το συζητήσουμε το στοιχείο αυτό και στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ashley Fox της ε, ομάδας ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις που έκαναν. Είναι εθνική αρμοδιότητα βεβαίως όλα αυτά. Άρα θα πρέπει να αναρωτηθούμε σε τι θα ωφελήσει η οδηγία, δηλαδή τι θα πρέπει να επιδιώκουμε. Ελπίζω ότι ο στόχος είναι να βελτιώσουμε τον αριθμό των προσώπων που καλύπτονται από τις συντάξεις, την ασφάλεια των συντάξεων, αλλά και να αυξήσουμε και τα χρήματα που λαμβάνουν όταν συνταξιοδοτούνται. Δηλαδή πάνω σε αυτά θα πρέπει να κρίνουμε την επιτυχία ή αποτυχία μας. Συμφωνώ με την κυρία Σέγκας που λέει ότι δεν θα πρέπει να εμείνουμε να έχουν επαγγελματικά προσόντα όλοι οι τραστείς γιατί αλλιώς βγάζουμε απ' έξω πολλούς ανθρώπους που θα έχουν σημαντικά πράγματα να συνεισφέρουν. Και νομίζω ότι έτσι αποκλείουμε και πολλούς συνδικαλιστές που για την ώρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των ε, συνταξιδοτικών αυτών ταμείων. Συμφωνώ με, τον, ε, με τους κύριους Στίφερμαν και Τσερούτη που λέει ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να προκαλέσουμε έξτρα κόστος και επιβάρυνση. Δεν χρειαζόμαστε κεφαλαιακές απαιτήσει. Δεν ξέρω πού προηγείται ο κ. Βαν Μέρτεν όταν λέει ότι χρειαζόμαστε ενοποιημένες απαιτήσει φερεγγιότητα για να αποφύγουμε και άλλε καταστροφές. Να με συγχωρείτε πολύ, αλλά ε, όπως τα λέτε εσείς, επίκειται άλλη καταστροφή για τους εργαζόμενους και για μείωση των συντάξεών του και για δυσκολία κάλυψής τους. Και μια ερώτηση για το πάνελ. Στην, ε, στο Ενωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία τα IAORP τα καθιδρύουν οι εργαζόμενοι. Ε, υποφελία των εργαζομένων τους, ίσως σε διαφορά με την Ολλανδία, όπου είναι ξεχωριστοί οργανισμοί τα IORP. Επομένως, πώς διασφαλίζουμε ότι οποιαδήποτε νέα νομοθεσία θα καλύψει όλη την ποικιλομορφία των IORP σε όλες τις χώρες μέλη και πώς εξασφαλίζουμε ότι θα αυξηθεί η προστασία χωρίς παραπέρα, παραπέρα συγγνώμη, κόστος διότι αν τα αποτελέσματα της οδηγίας οδηγήσουν τελικά σε μείωση του αριθμού των δικαιούχων, σε μείωση των συντάξεων που λαμβάνουν, τότε πραγματικά δεν βλέπω να υπάρχει ένας λόγος να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ασλή Φόξ. Για τους φιλελεύθερους τώρα. Η Σόφιν θέλετε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάλλον όλοι πολύ σύντομα μπορούμε να αποφασίσουμε για τους στόχους. Κανείς δεν θα έλεγε, μπα, ο στόχος μας πρέπει να είναι ένας διακανονισμός που να μειώνει τους δικαιούχους συντάξεων ή να είναι πιο και ότι αν περάσει οι συντάξεις. Όχι βέβαια. Αλλά το να ότι όλα είναι τέλεια τώρα και ότι αν περάσει νέα νομοθεσία θα τα χαλάσουμε όλα, δεν είναι ούτε αυτό αλήθεια. Άσυλη, δεν ξέρω τι γίνεται στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτοί που αποδυναμώνουν τα δικαιώματα των δικαιούχων στην Ολλανδία είναι ακριβώς τα στρατιωτικά ταμεία, γιατί δεν έχουν ασυλία από την οικονομική κρίση. Έχουμε ένα σταθερό σύστημα στις κάτω χώρες, αλλά όχι ότι είναι και απόλυτα ασφαλές. Έπειτα, για χρόνια τώρα προσπαθούμε να συζητήσουμε τις συντάξεις στην Ευρώπη. Και είναι σαν να απαγορεύεται η συζήτηση του θέματος. Μα αλλάζει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην αλλάζει, δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην αλλάζει ο τρόπος εργασίας, σαν να μην αλλάζει η αγορά εργασίας. Και αυτό το οποίο εμένα με ενοχλεί όλος είναι ότι πολλοί από αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις και λένε να μην αλλάξει τίποτα, να μείνουν όλα ως έχουν. Δεν μιλούν εκ μέρου των μελλοντικών συνταξιούχων. Είναι οι νέοι που επίσης δικαιούνται αξιοπρεπείς συντάξεις. Και αν δεν έχουμε εμείς τώρα το θάρρος να αναγνωρίσουμε ότι μπορεί να υπάρχουν αδυναμίες στο σύστημα, μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι, ε, τότε νομίζω ότι δεν είμαστε σωστοί απέναντι στους νέους. Και κύριε Στίβεμαν, συγγνώμη, ελπίζω να μην σας κατάλαβα καλά, αλλά άκουσα να λέτε ότι δεν χρειάζεται προστασία των καταναλωτών γιατί οι υπάλληλοι βασίζονται στους εργοδότες τους. Εγώ ελπίζω ότι μπορούν να βασίζονται στην νομοθεσία και στους νομοθέτες τους που θα διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, όχι στον εργοδότη τους. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να αντιγράψουμε τη Solvency 2 και για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, αλλά αν υπάρχουν κίνδυνοι, τότε ας σκεφτούμε τρόπους ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί. Αν δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά αν δεν υπήρχε κίνδυνος, δεν θα είμαστε εδώ να συζητάμε. Πρέπει επίσης να δούμε και το διασυνοριακό ζήτημα, γιατί αν δημιουργήσουμε μια πραγματικά ενιαία αγορά και αν πούμε ότι φτιάχνουμε αυτή την ενιαία αγορά και σε αυτό τον κλάδο, είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος αυτός. Τέλος. Ναι, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις διαφορές που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υιοθετήσουμε κανόνες που θα διασφαλίσουν τις συντάξεις όλων και των σημερινών συνταξιούχων αλλά και των αυριανών και μεθαυριανών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Σοφή. Εκ μέρους της Γκουέντζιαλ ο Μικέλ Ουρμπάν Κρέσπο έχει το λόγο. Δεν τον βλέπω όμως εδώ, λέει ο πρόεδρος. Α, εσείς εκ μέρους της Γκουέντζιαλ. Είμαι ο Μιγγέλ Ουρβέρ Κρέσπο της Γκουε, πρόεδρε. Ε, μπροστά μου είναι άλλο καρτελάκι, εντάξει, θέλετε σαν να είμαι εδώ πέρα αναπληρωματικό μέλος, αλλά δεν είμαι αναπληρωματικό, είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής αυτής. Δεν ε, ήμουν εδώ στην αρχή των παρεμβάσεων, γιατί είχαμε κάποια άλλη δραστηριότητα με άλλες οργανώσεις που φέραμε εδώ εκείνων που δεν έχουν ε, έγγραφα διαβίωση και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Πάντως το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα το σύστημα αυτό συντάξεων. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι, όπως το ξέρουμε και με άλλα παραδείγματα σε διάφορε χώρες. Πώ μπορούμε λοιπόν να διαχειριστούμε τα συστήματα συντάξεων, τα ιδιωτικά για να μην γίνονται τα λάθη που έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν γίνει, αλλά να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ευημερία τόσων <clears throat> που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτό που πάνω απ' όλα μας απασχολεί και το έχουμε πει εδώ και 20 μέρες η ασφάλεια που προσδίδουμε σε αυτές τις ιδιωτικές υπηρεσίες συνταξιοδότησης. Επίσης μας απασχολεί πολύ και το θέμα των επενδύσεων των Ιδρυμάτων αυτών συνταξιοδοτικών παροχών. Έχουμε διαπιστώσει ότι στη χώρα μου, για παράδειγμα, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα συστήματα προτιμησιακά και άλλα που έχει σαν αποτέλεσμα να χάσουν τις αποταμιεύσεις τους πάρα πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπόρεσαν δεν ε, είχαν τελικά την ασφάλεια που θέλανε με τις επενδύσεις των ε, Ιδρυμάτων αυτών. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει πάντα να είναι ένα συμπλήρωμα. Δεν θα πρέπει να καταργηθούν τα δημόσια συνταξιδιωτικά ταμεία και να αντικαταστηθούν πλήρως από τα ιδιωτικά. Επίσης, η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες πολλές επιχειρήσεις κάνουν τη διάκριση. Κάνουν διάκριση μεταξύ των εργαζομένων. Βάζουν διαβαθμίσεις. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα. Ο Σβέν και η έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Φυσικά και έχουμε διαφορετικά μοντέλα στις διάφορες χώρες μέλη και γι' αυτό δεν υπάρχει περιθώριο και δεν νομίζω κανείς να θέλει να αντικαταστήσει όλα αυτά τα συστήματα από ένα ενιαίο που να εξυπηρετεί όλους. Αλλά βέβαια, εδώ είναι σαν να έχουμε έναν ελέφαντα μέσα σε αυτό το δωμάτιο που δεν το κατονομάζουμε. Έχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια σήμερα και αμφισβητούμε κάποια μοντέλα τα οποία διασφαλίζουν τις συντάξεις που θα πρέπει να πληρωθούν. Το σύστημα το λογιστικό επιτρέπει ορισμένες χώρες να κρύβουν τις απώλειές τους. Ή τέλο πάντων να μην πω απώλειες, αυτήν την έλλειψη παροχών, την αδυναμία παροχών ε, για το μέλλον, εφόσον παραμείνουν χαμηλά τα επιτόκια. Τη συζήτηση αυτή θα την κάνουμε και για το πλαίσιο της οδηγίας Φερεγκαιότητα 2. Όμως αυτό το σύστημα, αυτό το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και για το κατά πόσο ένα σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει όλους ή όχι, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες πρέπει να δουν το εξή. Μήπω κάποιες επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν μεγάλο μέρος των κερδών του για να διασφαλίσουν τις μελλοντικέ συντάξεις αντί να επενδύουν για το μέλλον. Και δεύτερον, ακόμα κι αν τα συνταξιδοτικά ταμεία δεν είναι παραδοσιακοί οικονομικοί παράγοντες, μια μεγάλη τέτοια φούσκα θα μπορούσε να δημιουργήσει συστημικούς κινδύνους. Και γι' αυτό λοιπόν Χαίρομαι που βλέπω ότι όπα το σκέφτεται αυτό και δημοσιεύει και τα ποσά που διακυδεύονται εδώ. Στη Γερμανία ξέρω ότι οι εκτιμήσεις είναι 20-30 δις, ε, μείον δηλαδή στη δυνατότητα παροχών. Αλλού μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτερα ελλείμματα. Συνεπώς, ακόμα κι αν η εκθέση δεν καλύπτει τις κεφαλιακές απαιτήσεις, θα έπρεπε να μιλήσουμε και για αυτά τα ζητήματα και να ζητήσουμε από τους οικονομικούς επόπτες να το κοιτάξουν. Γιατί δεν μπορεί κανείς να πει δεν μιλήσαμε γιατί δεν θελήσαμε να πούμε για τον ελέφαντα που έχουμε μπροστά μας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον καθένα από τους τέσσερις ομιλητές. Πιστεύετε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στην ευρωπαϊκή οικονομία εξαιτίας της έλλειψης πρόβλεψης. Και αν ε, υπάρχει τέτοια υποπρόβλεψη, μπορείτε να μας δώσετε κάποια ποσά για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Γκίγκολ. Ένας ζητά ακόμα το λόγο, σαν catch the eye θα το πάρω και μετά θα επανέλθω στους στους τέσσερις ομιλητές μας. Και θα δούμε. Τόμας Μαν είναι ο επόμενος. Παρακαλώ. Κάτσε διάρκεια. Οι εμπειρογνώμονες κατέστησαν σαφές ότι υπάρχουν διαφορές στις χώρες μέλη, οι οποίες βεβαίως δεν είναι συμπτωματικές. Έχουν προκύψει από το διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο. Βεβαίως και το σύστημα των τριών πυλώνων δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες. Αυτά όλα πώς θα γίνουν ένα σύστημα. Δεν μπορούν. Η Σοφή Φανίν Φέλτ ήδη στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο είχαμε συζητήσει για το θέμα της δυνατότητας μεταφοράς. Κανένας δεν θέλει να φτιαχτούν τείχη. Αυτό που θέλουμε να επιτύχει είναι όπου υπάρχει αναγκαιότητα να καταργηθούν οι φραγμοί. Έχουμε διαφορές και είχαμε διαφορές στην στο όριο της ηλικίας εισόδου, πόσο ε, θα μείνουν τα χρήματα στις επιχειρήσεις, εάν θα είναι δυνατόν να καταβάλλονται οι συντάξεις εφόσον μετακινείται ένα πρόσωπο από μια χώρα μέλος σε άλλη. Ε, δηλαδή έχουμε ήδη επιτύχει σημαντικό βαθμό ευκαμψίας. Δεν βλέπω πουθενά να κρύβεται κανένα θέμα ταμπού. Και πέρα από αυτό, ορισμένοι, στην χώρα μου τουλάχιστον, απέδειξε το σύστημα ότι είναι ασφαλές απέναντι σε οποιασδήποτε περιπτώσεις αφαιρεγγιότητας. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι επίσης σαφές. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Πρόκειται για μια κοινωνική διάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλά ένα χρηματοδοτικό προϊόν μεταξύ πολλών. Και αυτό κατέστησε σαφές. Αυτό σημαίνει όμως ότι Πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτά τα επιχειρήματα περί Solvency 2. Δεν έχει καμιά σχέση με τη Solvency 2. Ο Σβέν Κίγκολ που μίλησε πριν έχει δίκιο. Το ερώτημα είναι πώς μπορούν να διατηρηθούν όρθια τα συνταξιωτικά αυτά συστήματα εν ώψη της πολιτικής πολύ χαμηλών επιτοκίων τη Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό πρέπει να το αναλλάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να καλύψει κανείς. Βεβαίως και προβληματίζει πολλούς. Αυτές οι επαγγελματικέ συντάξεις θα διατηρηθούν εφόσον δεν έχουν απόδοση για την ώρα. Ορισμένοι θέλουν να τι εγκαταλείψουν. Αυτή θα ήταν και η χειρότερη δυνατή εξέλιξη ωστόσο, διότι υπάρχει ένα ξεχωριστό benefit στην, ε, μέσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα και αυτό θα πρέπει να παραμείνει. Τώρα, Holistic Balance Sheet. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ΑΕΟΠΑ έχει θέσει ερωτήσεις και προς τους τέσσερις πανελίστ 111 ερωτήσεις για την περαιτέρω εργασία για την ε, ΑΙΟΠΑ. Κατά πόσον έχετε απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές και απέφερε κάτι η προσπάθεια αυτή. Δεύτερο, οι ρήτρες εξουσιοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί εξουσιοδότηση και από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπει μέσα και μια κατεξουσιοδότηση πράξη ώστε να μπει εκεί ο αξιολόγηση του κινδύνου. Τέλος, η ρήτρα αναθεώρησης. Εκ παραλλήλου έχουμε απόφαση τη οικονομική επιτροπή και τη επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί το ίδιο πράγμα συζητείται και λαμβάνεται απόφαση και στην Επιτροπή απασχόληση για το θέμα τη αναθεώρηση δεν είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά αν θα γίνει αναθεώρηση σε 4 ή σε 6 χρόνια. Η Επιτροπή Απασχόληση θέλει 6 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει 4 χρόνια. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση προ όλου, όλα τα μέλη του πάνελ. Ευχαριστώ. Βρίσκω ότι η συζήτηση αυτή έχει οδηγήσει και σε μια συνειδητοποίηση και από πλευρά συναδέλφων που δεν είχαν προσέξει τόσο πολύ το θέμα. Μάλιστα, πολλέ ερωτήσει για τα μέλη του πάνελ, βεβαίω λίγο χρόνο. Εμείς έχουμε συνηθίσει να δρούμε έτσι, το ίδιο όμως θα ζητήσουμε τώρα και από σας. Η κυρία Σέγκαρς. Σας ευχαριστώ. Ε, ρωτήσατε κύριε Τάγκα αν ε, είναι ευπρόσδεκτη μια οδηγία ε, και αν κάτι θα βελτιώσει. Ε, ναι, είναι ευπρόσδεκτη γιατί ο κόσμος αλλάζει και αυτό είναι απάντηση και προς την κυρία Ιντφέλτ η νομοθεσία οφείλει να ανταποκρίνεται και να αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές. Είτε είναι αυτές οι αλλαγές ε, στα προγράμματα, είτε είναι στη δημογραφία, είτε είναι ε, νομοθετικές ε, αλλαγές. Έτσι πρέπει να αλλάξουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος σήμερα που μπαίνει στην αγορά εργασίας να μπορεί να αναμένει μια καλή σύνταξη αύριο μεθαύριο. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία λοιπόν που μπορεί να κάνει η οδηγία αυτή και να εναμφύρει καθώς και να διαδώσει την καλύτερη πρακτική ιδιαίτερα όσον αφορά την διακυβέρνηση. Ε, συμφωνώ επίσης με την ανάλυση του κυρίου Φόξ όσον αφορά την επιτυχία, ότι δηλαδή ο κόσμος θα εξοικονομεί περισσότερο για την σύνταξή του. Ρώτησε αυτό το θέμα της ε, διαφορετικότητας και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αναγνωριστεί το θέμα αυτό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά δηλαδή τις ε, περισυντάξεων ε, διατάξεις. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ισχύουν κάποιε ελάχιστε προδιαγραφέ, αλλά να μπορούν ταυτόχρονα να αναγνωρίζονται οι εθνικέ ιδιαιτερότητε. διότι οι περί συντάξεων διατάξεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μάλιστα κατά πολύ. Πρέπει ωστόσο να εξασφαλίσουμε μια νομοθεσία που θα ανταποκρίνεται στο σκοπό αλλά και, θα, και στο κοινό στόχο ότι δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα παροχής επαγγελματικής σύνταξης ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πω ότι δεν βλέπω το θέμα της ε, ρυθμιστικής διαιτησίας με τον ίδιο τρόπο όπως ε, το βλέπει η ΕΙΟΠΑ. Τώρα, ε, αυτό που είπα ότι ο κόσμος αλλάζει, αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε πολύ μεγάλες δημογραφικές μετακινήσεις όπου, όπου θα έχουμε το ποσοστό που θα εξαρτάται από την σύνταξη να διπλασιάζεται και πολλοί κόσμος θα μείνει εκτός ε, τέτοιων διατάξεων. Όταν βλέπουμε λοιπόν το πλαίσιο, θα πρέπει να μας ανησυχήσει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν μη επιθυμητές συνέπειες και άρα λοιπόν ε, ε, το αποτέλεσμα να μην είναι λιγότερη σύνταξη οδοτημένη. Έτσι όπως έχει τώρα η οδηγία ε, θα σήμαινε πολύ μεγάλο παραπανήσιο κόστος. Δηλαδή στη χώρα μου 220 δις λίρες ε, θα επιβάρυνε τα συνταξιδοτικά ταμεία. Οπότε η αντίδραση των εργοδοτών θα ήταν να τα σταματήσουν. Και αυτό θα ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε συμβεί. Και εγώ συμφωνώ όπως είπε ο κύριος Μάν και εγώ συμφωνώ μαζί του απόλυτα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εξαπλωθεί το, η παροχή συντάξεων και διασυνοριακά όπου αυτό γίνεται. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των μακροπρόθεσμων χαμηλών επιτεκίων. Υπόθηκε ότι οι σημερινές ε, λογιστικές προδιαγραφέ κρύβουν το πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι πολύ βεβαία όταν το συζητάμε αυτό στην Pensions Europe αλλά και στην Εθνική μας Ένωση ε, των Σταξιδικών Ταμείων. Είναι το θέμα το οποίο απασχολεί τα ταμεία αυτή τη στιγμή και κρατάει ξύπνιο τον κόσμο που ασχολείται με αυτό. Θα πρέπει επίση να δούμε μήπως αυτή η αφαιρεγγιότητα 2 κάνει χειρότερα τα πράγματα. Μήπω τυχόν δηλαδή οθήσει τον κόσμο στο να επενδύσει στα χαμηλής απόδοσης ε, δεξιτικά ε, ταμεία ε, αντί να επενδύσει σε άλλα πιο κερδοφόρα. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα διατηρήσουμε κάποιες αρχές, ότι θα πιέσουμε και θα αυξήσουμε την, τις προδιαγραφές διακυβέρνησης αλλά και τις επικοινωνίες μας για τρόπο που να είναι ωφέλιμος και για τα κρατημέλη και για τα ταμεία, ε, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές συνθήκες και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους παρέχονται οι συντάξεις στην Ένωση, με στόχο πάντοτε την διάδοση της ε, καλής ποιότητας συνταξιδοτικών ταμείων και κάλυψης, συνταξιδοτικής κάλυψης. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μέρτενα. Εγώ θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις, ερώτηση, τις ερωτήσεις και να απαντήσω με δύο παρατηρήσεις. Δεν νομίζω ότι η Solvency 2 για τις IOP θα καταστεί αναγκαία. Ούτε και εγώ υπέρ αυτής. Αυτό που ζητώ είναι οι κεφαλαϊκές απαιτήσεις να είναι πιο εναρμονισμένες με τρόπο που να αποφεύγεται ε, το ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Βλέπουμε ωστόσο συνταξιωτικά ταμεία τα οποία μετακινούνται στο Βέλγιο. Περιορισμένα σε αριθμό, ωστόσο όλο και περισσότερο. Και κυρίως λόγω των επιτοκίων που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτό παρατηρώ εν πάση περιπτώσει. Δεύτερο, βλέπω ότι οι κεφαλαϊκές απαιτήσει που μας έχουν επιβληθεί αν θέλετε έτσι, ε, τέλος πάντων επιβάλλονται ούτως ή άλλως είτε μέσω της εργασίας της ΑΙΟΠΑ ή από άλλους οργανισμούς. Καλύτερα θα ήταν να ρυθμιστούν τα πράγματα αυτά στην ίδια την οδηγία αντί να χρησιμοποιούνται άλλων ειδών μηχανισμοί για να μπουν απαιτήσει ε, φερεγιότητα που να είναι και χειρότερες. Αν λύσετε τα προβλήματα αυτά στο επίπεδο της οδηγίας, τότε μπορείτε να επηρεάσετε τη ρύθμιση αυτών των παραμέτρων. Αν δεν τα ρυθμίσετε, τότε δεν μπορείτε και να τις επηρεάσετε. Ο λόγος για τον οποίο αναφέρθηκα στην ε, ε, Solvency 2, δεν είναι επειδή μου αρέσει τόσο πολύ, αλλά επειδή περιλαμβάνει και πρόβλεψη για διαμεθοριακή δραστηριότητα. Και εδώ απαντώ στον κύριο Τάγκ. Η απάντηση θα πρέπει να είναι ότι ορισμένες IOP θα πρέπει να είναι διαμεθοριακές και άλλες όχι. Όπως γνωρίζουμε, το δικαστήριο ερμηνεύει ευρέως ως διαμεθοριακή ε, δραστηριότητα. Ακόμα και ενδοεπικρατειακές, ας πούμε, δραστηριότητες οι απαιτήσει τη οδηγία εφαρμόζονται μόνο σε συνταξιωτικά ταμεία τα οποία βρουν διαμεθοριακά, δηλαδή τα οποία για παράδειγμα μετακινούνται και μετεγκαθίστανται στο Βέλγιο. Εκεί πρέπει να ε, ρυθμιστεί το επίπεδο της ε, αλληλεγγύη. Εάν τα συνταξιωτικά ταμεία είναι αλληλέγγυα κατά κάποιο τρόπο, τότε δεν είναι διαμεθοριακά, λειτουργούν μέσα στην μεθόριο και οι απαιτήσει που περιλαμβάνουν στην οδηγία δεν εφαρμόζονται ένα προ ένα. Αυτά που είναι όμως που δραστηριοποιούνται διαμεθοριακά θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στίφερμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρκετές ερωτήσεις βέβαια. Ας αρχίσω με μια διευκρίνηση που ανέφερε η κυρία Ιντφέλτ. Όταν μιλώ για προστασία καταναλωτών ως αυτή αντιτίθεται στο εργασιακό δίκαιο ενώ ότι αυτά που κινούνται μέσα στα πλαίσια του εργασιακού δικαίου που καθιδρεί το πλαίσιο τουλάχιστον στη Γερμανία αλλά πόσο γνωρίζω και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το δίκαιο της εργασίας δίνει στον εργοδότη μια καλύτερη θέση από ότι θα έδινε σε αυτόν σε αυτήν το δίκαιο προστασία των καταναλωτών. Και στη Γερμανία, λόγω της άμεσης σχέσης μέσα σε αυτό το τρίγωνο του εργοδότη εργαζόμενου και στην περίπτωση αυτή της IORP ή Group Insurance ή οτιδήποτε άλλο, η νομική κατάσταση και ο νομικός σύνδεσμος είναι μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δεν προστατεύεται. Αν εξετάσετε προσεκτικά τη γερμανική κατάσταση θα δείτε ότι ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοι προστατεύεται καλύτερα σε αυτή την άμεση από ό,τι θα ήταν προστατευόμενο σε μια άμεση σχέση με μια ασφαλιστική εταιρεία. Ο Σβέν Γκίγκολτ αναφέρθηκε σε ορισμένους αριθμούς σε σχέση με την έλλειψη προβλέψεων στα συστήματα της Γερμανίας. Τα νούμερα που ακούγονται συχνά στον τύπο δεν έχουν τη σωστή προοπτική των επαγγελματικών συντάξεων στη Γερμανία. Οι οποίε επαγγελματικέ συντάξει στη Γερμανία, τουλάχιστον να εξετάσετε τα στοιχεία του ενεργητικού, τουλάχιστον οι μισέ από αυτέ περίπου δηλαδή 270 με 280 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι σε book reserves. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σε αποθεματικά βιβλία δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν εξετάσετε από μια προοπτική διεθνή ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστά στοιχεία ενεργητικού των συντάξεων. Τα χρήματα βρίσκονται μέσα στην επιχείρηση και στη Γερμανία είναι προστατευμένα πολύ καλά τα χρήματα αυτά, διότι αυτό το σύστημα των αποθεματικών βιβλίων υποστηρίζεται από 94.000 Γερμανούς εργοδότες όλων των μεγεθών και όλων των οικονομικών κλάδων. Είναι αυτή η, το γερμανικό σύστημα προστασίας κατά της αφαιρεγγιότητας και με ένα ιστορικό 40 ετών στο πεδίο της προστασίας καθένας αφαιρεγγιότητας, εγώ δεν αισθάνομαι δυσάρεστα με αυτή την κατάσταση όπου έχουμε book reserves και όπου θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη προβλέψεων. Εκεί όπου τα, αισθήματά μας, τα συναισθήματά μας είναι ανάμεικτα και ίσως μάλιστα και πιο αρνητικά, είναι η παρούσα κατάσταση των επιτοκίων που όντως αντιμετωπίζουμε τώρα, όπου επιχειρήσεις αναγκάζονται να αποθεματοποιούν πολλά, περισσότερα χρήματα, να βάζουν δηλαδή σε αυτά τα αποθεματικά βιβλία λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων. Ο κ. Μαν ε, εξεδίδωσε και αυτός ανάμεικτα συναισθήματα σχετικά με την HBS. Και εγώ δεν ξέρω αν η HBS σημαίνει ένα σύμβολο για την Solvency 2, ένα είδος Solvency 2 Light. Και πάντως δεν είναι κάτι που εγώ θεωρώ σημαντικό. Να υπάρχει ένα καθεστώς δηλαδή το οποίο να ρυθμίζει τα των επαγγελματικών συντάξεων μέσα στην ποικιλομορφία του Δεν είναι ένα είδος ασφαλιστικής εταιρεία οι επαγγελματικέ συντάξει, είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, όπου εμείς στη Γερμανία λέμε συνταξιωτικά ταμεία, ΑΙΟΠ, έχουν μια ιστορία 170 ετών και είμαι βέβαιο ότι όσον οι επαγγελματικέ συντάξει στη Γερμανία είναι εθελοντικές αν βάλουμε κάτι όπως η Solvency 2 για τα IOPS, οι επιχειρήσει δεν θα δίνουν πλέον υποσχέσεις που να καλύπτονται από IOPS. Στη Γερμανία υπάρχουν διάφοροι τρόποι που ε, υπόσχονται τα δικαιώματα των συνταξιοδοτημένων οι επιχειρήσεις, αλλά είναι Εθελοντικέ, Από την άποψη του εργοδότου, ωστόσο, είναι κόστος, είναι επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και όπως όλες οι επενδύσεις ελέγχονται και αν υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι επενδύσεων στον ίδιο τομέα με το ίδιο αποτέλεσμα, ο επιχειρηματίας μπορεί να διαλέξει τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε εδώ πάρα πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αλλά όλοι πρέπει να έχουν τον ίδιο χρόνο, όπως καταλαβαίνετε. Ο κύριος Τσερούτη, τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Υπάρχει βέβαια μια ευρωπαϊκή διάσταση, εννοείται, και αρχίζει από τη δημογραφική εικόνα που έχουμε. Και το διαπιστώσαμε από αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα. 75 εκατομμύρια πρόκειται να σταξιδοτηθούν μέχρι το 2020 και αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλος ο αριθμός. Κάπου 220 εκατομμύρια είναι ήδη τώρα. Καταλαβαίνετε ότι η τάση είναι πολύ μεγάλη. Είναι μια τάση που έχουμε τα τελευταία χρόνια και η οποία μας οδηγεί να βάλουμε το συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια έκτακτη κατάσταση. Η Ευρώπη, λοιπόν, πρέπει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και τα συστήματα τα οποία διαθέτει να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Άρα τα κεφάλαια, τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν τα ταμεία επαγγελματικών συντάξεων μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Όντω, η πρόταση Επιτροπή περιλαμβάνει διάφορε βελτιώσει όσον αφορά του επενδυτικού κανόνε για να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία σε περισσότερα προϊόντα κλπ. Τώρα, στρεφόμενοι προς το μέλλον. Όσον αφορά τους ενδυνάμει κινδύνους οι επαγγελματικέ συντάξεις σίγουρα είναι ένα μέρος της λύσης για να προσφέρουν ε, περισσότερη ασφάλεια σε όσους τις προτιμούν. Οι κίνδυνοι θα ήταν μεγαλύτεροι αν δεν υπήρχε αυτή η αναλλακτική. Βέβαια πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία. Τι πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την αναθεώρηση της οδηγίας αυτής και τι είναι αυτό που παραμένει αρμοδιότητα των χωρών μελών. Τίποτα άλλο. Και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Ο Πρόεδρος. Ωραία. Μπράιεν, άκουσες πάρα πολλά. Οπότε τώρα. Εσύ μπορείς να καταλήξεις τα πρώτα σου συμπεράσματα και να προχωρήσεις μετά στην εκπόνηση της εκθεσής σου. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πράγματι. Θα χρειαστώ βέβαια ειδικέ ιδιότητες για να μπορέσω όλα αυτά να τα συγκεντρώσω. Πάντως είμαι ευγνώμων και στους τέσσερις ομιλητές μας που ήρθαν και με τόση σαφήνεια απάντησαν στις ερωτήσεις των συναδέρφων. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων επίσης όλους τους συναδέρφους και τους σκιώδες, αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας που ήρθαν σήμερα και έθεσαν τις ερωτήσεις τους. Πολύ βασικός πρώτη αρχή να πούμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τα χρήματα κάποιου άλλου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη στους ώμους μας, σε εμά, που πολύ σωστά θέλουμε να ενημερώσουμε τους όρους της οδηγίας αυτής που είναι παλιά, ε, είναι 13 ετών περίπου και να την διαμορφώσουμε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές καταστάσεις. Πρέπει να το κάνουμε με αναλογικότητα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εθελοντικά μέρος του μισθού τους, του εισοδήματός του, μηνιαίου, τα κτλ. να το επενδύσουν εκεί. Ο στόχος βέβαια είναι κάποια στιγμή στο μέλλον να έχουν σύνταξη από τα χρήματα αυτά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη απόφαση που παίρνει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, που στηρίζουν έτσι το σύστημα επαγγελματικών συντάξεων που υπάρχει σε διάφορες χώρες. Συγχρόνως βέβαια πρέπει να ενθαρρύνουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, εργοδότες, να μπουν σε τέτοια συστήματα και να έχουμε και ένα σύστημα που να είναι δίκαιο για όλους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να καταλάβουμε επίσης ότι οι μεγάλες αλλαγές που γίνονται όσον αφορά ε, τις ε, διαφορές επίσης μεταξύ των μεθόδων που έχουν να κάνουν ε, με τα κέρδη της συντάξης της εγκυμένης και τις μη εγκυμένης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας λοιπόν το εξή ότι γενικά μιλώντας, ναι, είμαστε υπέρ της πρότασης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γενικά. Βέβαια, έχει τροποποιηθεί μετά από τις ειδήσεις που έγιναν στο Συμβούλιο. Η γενική αναγνώριση πάντως είναι ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να προχωρήσει. Ήμουνα εθνικός βουλευτής 16 χρόνια και σε κάθε νομοθέτημα που πέρναγε από το Ελλαδικό Κοινοβούλιο, που είναι σαν και αυτό. Αν έχετε ένα νομοθέτημα 13-14 ετών, έτσι κι αλλιώς πρέπει να το βάλεις κάτω, να το ξαναδείς, να το εξυγχρονίσεις και να βεβαιωθείς ότι τα επιχειρήματα τα οποία οδήγησαν σε αυτό ισχύουν ακόμα ή δεν ισχύουν οπότε πρέπει να το αλλάξεις. Αυτό κάνουμε και εδώ τώρα. Οπότε γενικά μιλώντας, ναι, είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση της Επιτροπής. Δεύτερον, με πολύ ενδιαφέρον άκουσα από όλου ουσιαστικά τους ομιλητές το βασικό επιχείρημα για να έρθουν οι φραγμοί όσον αφορά τα διασυνοριακά ιδρύματα συνταξιδοτικών παροχών. Και μίλησαν υπέρ διασυνοριακών τέτοιων ιδρυμάτων. Αν εμεί θέλουμε περισσότερα τέτοια στο μέλλον, μόνο 86 έχουμε τώρα από το 2003. Είναι πολύ λίγα αν σκεφτούμε πόσε είναι οι χώρε μα. Αν λοιπόν είμαστε σοβαροί και πράγματι θέλουμε περισσότερα διασυνοριακά ιδρύματα εξωτερικών παροχών στο μέλλον, τότε πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι φραγμοί. Γιατί δηλαδή δεν έχουμε περισσότερα. Αυτό το πρόβλημα να εντοπίσουμε. Ποια είναι τα εμπόδια. Αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν στα πλαίσια των συζητησιών μας. Και τρίτον, φυσικά και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Αντί λοιπόν την νομοθεσία αυτή να τη δούμε σαν κάτι που επιβάλλεται στις χώρες μέλη, πρέπει να πούμε ότι θέλουμε να έχουμε έναν βασικό στόχο προστασίας παντού σε όλες τις χώρες μέλη. Αν το κάνουμε αυτό, τότε συγχρόνως πρέπει να αφήσουμε τις χώρες να το διαχειριστούν όπως νομίζουν και να αφήσουμε όποιες χώρες θέλουν να συμπεριληφθούν με τον τρόπο που θέλουν. Και τέταρτον, κάτι που είπανε πολλοί συνάδελφοι. Προσπαθούμε να ελεγχιστοποιήσουμε το κόστος. Μα μιλάμε για ένα κλάδο και άκουσα αυτά που είπε ο κ. Γκίγκολτ για τον ελέφαντα στην αίθουσα. Όντως, ζούμε σε ένα περιβάλλον πολύ χαμηλών επιτοκίων και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην επιβάλλουμε επιπλέον κόστος ούτε στους εργαζόμενους ούτε στα ιδρύματα αυτά. Συμφωνώ με του συναδέλφους που είπαν ότι ο κόσμος αλλάζει δημογραφικά, οι πρακτικές εργασίας είναι αναπόφευκτο. Όλο και περισσότεροι πολίτες μας θα ταξιδεύουν και θα βρίσκουν δουλειά σε άλλες χώρες από τις δικές τους. Και όσο ταξιδεύουν θα χρειάζονται διαφορετική σταξιδιωτική κάλυψη, γιατί υπάρχουν διαφορετικά σταξιδιωτικά προγράμματα, οπότε πρέπει να εξυγχρονίσουμε το σύστημά μας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί που πολύ σωστά ταξιδεύουν και αλλάζουν χώρους εργασίας να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Και τέλος πρέπει να συζητήσουμε, το είπε και τον ρόλο των ταξιδιωτικών επαγγελματικών ταμείων όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και πώς θα λειτουργεί καλά η αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χρήματα τα οποία περιμένουν να επενδυθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φροντίσουμε ότι γίνεται σε ένα μέρος να μην επηρεάζει αρνητικά κάτι που γίνεται σε κάποιο άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και την πρόταση του Επιτρόπου Τίλεμανς για την καλύτερη νομοθέτηση, καλύτερη νομοθετική ρύθμιση. Να την έχουμε στο μυαλό μας τη συζήτηση αυτή που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε μη ρεαλιστικές λύσεις. Και το λέω αυτό και για αυτή την πρόταση. Πάντως όσον αφορά εμένα πιστεύω ότι η συζήτηση που είχαμε σήμερα ήταν πλήρης και χαίρομαι που το θέμα των απαιτήσεων Θερακιότητας 2 αναλύθηκε από τους συναδέρφους. Δεν, δεν υπάρχει στήριξη να συμπεριληφθεί η απέτηση αυτή. Οπότε καλώς βγήκε. Πάντως, όσα είπαν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση σήμερα είναι ότι χρειάζεται ε, ρύθμιση, χρειάζεται αναθεώρηση, χρειάζεται δικαιοσύνη και πρέπει σωστά να νομοθετήσουμε. Ελπίζω λοιπόν στην έκθεσή μου που θα είναι έτοιμη πριν το καλοκαίρι να αντικατοπτρίζονται όλες αυτές οι ιδέες. Και από εκεί και πέρα προσβλέπω στη στήριξη των συναδέρφων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ακρόαση, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος Φέρμπερ, Ευχαριστούμε θαυμάσια. Σύνοψη ευχαριστώ και τους τέσσερις ομιλητές που έλαβαν μέρος στην ακρόασή μας και βεβαίως ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας στη μελέτη του θέματος και θα παρακολουθούμε και θα παρακολουθείτε και εσείς το έργο μας. Είμαστε διαφανείς, απόλυτα διαφανείς και ο καθένας μπορεί να παρακολουθεί το τι πράττουμε. Χαίρομαι διότι ε, είμαστε πάντοτε μέσα στα χρονικά πλαίσια των εργασιών μας γιατί έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα. Είναι το υπαριθμό 4 τώρα, έλεγχος των κατεξουσιοδότησης συμπράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. Όταν δηλαδή ήδη έχουμε εγκρίνει τη σχετική νομοθεσία, μήνες πολλούς ή και χρόνια μετά ε, συζητούμε τα θέματα αυτά. Έχουμε τον κύριο Μάριο Νάρα τη Γενικής Διεύθυνσης ΦΙΣΜΑ. Καλώς ήρθατε στην ε, συνεδρίασή μας και από την ΑΙΟΠΑ Justin Reid, επικεφαλής της Ενότητας Πολιτικής και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 Okay, scrutiny slots is only for those who like it. <laughs> That's what I learned now. So, it's already our seventh. Η έβδομη μηνιαία εξέταση των ε, κατεξουσιοδότησης πράξεων και εκτελεστικών μέτρων των εποπτικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδίδουμε μεγάλη σημασία την ε, ορθή εκτέλεση αυτών των ελέγχων. Έχουμε κάνει και άλλες ανταλλαγές απόψεων από το περασμένο φθινόπωρο και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε τακτικά στις συναντήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και ως γνωρίζετε κατεξιότητες συμπράξεις και εκτελεστικά μέτρα είναι πολλά και συχνά το περιεχόμενό τους είναι πολύ τεχνικό. Παρ' όλα αυτά έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλές από τις πράξεις αυτές και θεωρούμε ότι η συζήτηση που γίνεται και στο κοινό είναι από τα θέματα κοινά που απασχολούν πάρα πολύ το κοινό. Θα ασχοληθούμε τώρα με ιδιαίτερα ε, ειδικά μέτρα ε, της οδηγίας Solvency 2 και ήδη από να το καλώς ορίσατε στον κύριο Μάριο Νάβα, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΦΙΣΜΑ, καθώς και τον ε, τριματάρχη της ΑΙΟΠΑ μέτρα λοιπόν θα εγκριθούν υπό την μορφή κατεξουσιοδότηση πράξεων και η πρώτη αυτή νομοθεσία θα καλύψει πλήρη ισοδυναμία για την Ελβετία και προσωρική, προσωρινή ισοδυναμία για Αυστραλία, Βερμούδα, ε, ε, Βραζιλία, Καναδά, Μεξικό και Ενωμένες Πολιτείες. Η ΑΙΟΠΑ έχει δώσει τεχνικές συμβουλές ήδη από τον Ιανουάριο 2015 αυτές οι ισοδυναμίες πρόκειται να εγκριθούν όπου να είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες πράξεις μετά από τις θερινές διακοπές. Πράξεις ισοδυναμίας θα πρέπει να παρουσιάζονται αναχώρα και ανα ε, τομέα μέσα στα πλαίσια των σχετικών οδηγιών αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Τώρα σας προσκαλώ λοιπόν τους κυρίους ε, Νάβα και ε, τον ε, Ματάκη της ΑΙΟΠΑ να προχωρήσουμε σε ανταλλαγή απόψεων. Ποιος θα αρχίσει, η ΑΙΟΠΑ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει, θέλετε να αποφασίσω. Αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Μάριο. Καλά λοιπόν, αν θέλετε να δώσετε την, το μικρόφωνο πρώτα στον άλλο, δεν έχω αντίρρηση. Έφυγε ο μπραιαν Hayes βέβαια, αλλά Με μεγάλη χαρά άκουσα τη συζήτησή σας για τα IRP και τις συντάξεις. Όπως γνωρίζετε είναι ένας ακόμη από τους τομείς όπου η μονάδα μου και εγώ προσωπικώς έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μου φάνηκε η συζήτησή σας πάρα πολύ διαφωτιστική. Και ευχαρίστω θα συνεργαστούμε μαζί σας και στο προσεχές μέλλον. Τώρα, τούτου λεχθέντος, θα αρχίσω με μια σύντομη εξήγηση. Υπάρχουν τρεις νομικές βάσεις όπως είπατε τρεις νομικές βάσεις για την ισοδυναμία. Ισοδυναμία για ευρωπαϊκές ασφαλιστικές με θηγατρικές σε τρίτες χώρες, άλλες με θηγατρικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ισοδυναμία για την αντασφάλιση. Είπατε ήδη και σωστά ότι υπάρχουν δύο νομοθετικές πράξεις στον αγωγό, μία που δίνει πλήρη ισοδυναμία στην Ελβετία και η άλλη που δίνει προσωρινή ισοδυναμία, προσωρινή δηλαδή 10 ετών στις χώρες που αναφέρατε, δηλαδή Αυστραλία, Βερμούδα, Καναδά, Μεξικό και Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης σωστά είπατε ότι οι εκθέσεις μας, οι αποφάσεις μάλλον περί ισοδυναμίας βασίζονται σε εκθέσεις της ΑΕΟΠΑ, βασίζονται σε αυτές, έτσι. Επομένως λαμβάνουμε τις ...εκθέσει της ΑΙΟΠΑ ως σημείο αφετηρίας, αλλά οι πράξεις είναι δική μας απόφαση. Έχουμε ένα δεύτερο κύμα τώρα αποφάσεων ισοδυναμίας για το φθινόπωρο του 2015. Το πεδίο εφαρμογής δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Με ρωτήσατε για την αποδέσμευση αναχώρα, unbundling δηλαδή και ανανομική βάση. Πιστεύω ότι ο Επίτροπος ήδη είπε ότι καταρχήν είναι υπέρ της ε, απόψεως αυτής και βεβαίως και εγώ το ίδιο τότε ε, είμαι λίαν υπέρ της δυνατότητας αυτής. Σας ευχαριστώ βεβαίως για την προσοχή που δίνετε στο θέμα. Είχα την τύχη να είμαι μαζί με τους κυρίους Μπουρκαρντ Μπάλτ, και άλλους όταν συζητούσαμε τη σκοτεινή εκείνη νύχτα του Νοέμβρη 2013 νομίζω ήταν. Ο Ιβο Μπέλετ ήταν επίσης παρόν. Θυμούμε ο Μπορκάρτ. ήταν ο ήρωας της νύχτας εκείνης. Ε, μακρά νύχτα εκείνη και ειδικά για τη συζήτηση αυτή το, της ισοδυναμίας. Καταφέραμε να επιτύχουμε ο Κρίς Σκίνερ ήταν επίσης παρόν. Αυτό που ακόμη εξακολουθώ να θεωρώ ήδη 1,5 χρόνο μετά, μια συμβαστική λύση ήταν πολύ ισορροπημένη για τις ξεκάθαρες υποθέσεις ισοδυναμίας και για τις άλλες που ήταν ας πούμε work in progress, δηλαδή προχωρούμε προς την πλήρη ισοδυναμία. Άρα βρισκόμαστε τώρα στην προσωρινή ισοδυναμία. Άρα είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δίνετε και ο Επίτροπός μου σημειώνει τα όσα είπατε για την αποδέσμευση ανά χώρα και ανά τομέα και είμαστε ε, ε, πολύ θετικοί απέναντι σε αυτό. Υπάρχει και η ανάγκη να υπάρξει μια ισορροπία σε ό,τι αφορά την μείωση του αριθμού των νομοθετικών πράξεων και να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Μάριο. Δεν θέλω να ακούσω όλες τις περίεργες λεπτομέρειες της σκοτεινής εκείνης νύχτας. Δέχομαι αυτά που είπατε. Ο κύριος Ρέι έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Πριν περάσω στις αντιστοιχίες, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να έρθω εδώ. Άκουσα τα όσα συζητήσατε για τις ε, συντάξεις και όπως καταλαβαίνετε και εμείς η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων ενδιαφέρεται όλος ιδιαίτερος. Θέλουμε οι ρυθμίσεις να ωφελούν και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ασφάλισης και κατασφάλισης και εκείνες των τρίτων χωρών. Θέλουμε συγχρόνως βέβαια να υπάρχει επαρκής προστασία. Η σημασία που έχει απόφαση αυτή αντιστοιχίας είναι μεγάλη Συζητάμε λοιπόν για τη συνεισφορά τώρα του ΕΟΠΗ. Εδώ θέλω να αναφερθώ στις διάφορες εκτιμήσεις που έκανε η ΕΟΠΑ, την αξιολόγηση δηλαδή, και επαναλάβω και εγώ αυτό που ακούσαμε πριν, ότι η συμβουλή και η ανάλυση είναι το σημείο κίνησης για αποφάσεις εξουσιοδότηση πράξεων. Όσον αφορά την πλήρη αντιστοιχεία, όσον αφορά την Ελβετία, τις Δεσμούδες και την Ιαπωνία. Έγινε ανάλυση της νομοθεσίας των χωρών αυτών, η εποπτική τους νομοθεσία και η πρακτική, οι διαβουλεύσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΗ. Όσον αφορά τώρα τις άλλες χώρες, ο Καναδάς, Μεξικό, Βραζιλία κτλ. Ο στόχος μας ήταν να έχουμε έτσι μια βάση για συζήτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τρίτες χώρες όσον αφορά την αντιστοιχία αυτή. Υιοθετήσαμε μια διαφορετική προσέγγιση. Εξετάσαμε τα εποπτικά καθεστώτα των χωρών αυτών και τα συγκρίναμε με τα δικά μας. Γι' αυτό και αποφασίσαμε για ένα προσωρινό καθεστώς αντιστοιχίας βάση του 2.2.7. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής μας. Τώρα. Ή εισηγητή μάλλον. Κάθριν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκπρόσωπο του ΕΙΟΠΑ. Όσον αφορά την αντιστοιχία με τρίτες χώρες, ο λόγος που το έχουμε αυτό για τις πιστώσεις και αφαιρεγγιότητα είναι για να μην υπάρχουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα. Και θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επιτροπό Γήλολος ιδιαίτερο, ο οποίο στην επιστολή του έλεγε ότι θα εγκριθούν τα μέτρα αυτά όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θέλω, μια που έχω την ευκαιρία εδώ, να επαναλάβω ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε αυτό και ότι είναι καλό μεμονωμένα να εξετάζουμε τις διάφορες περιπτώσεις και να μην τις ομαδοποιούμε, γιατί τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυσκολεύεται περισσότερο. Εάν δεν συμμορφωθεί με αυτές τις ε, ταξιοσχεδότηση αντιστοιχίες, θα υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τα κεφάλαια και θα δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα, κάτι το οποίο κανείς μας δεν θέλει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως θα να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τι μπορούμε να περιμένουμε με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις αυτές. Θέματα βάσει πάντα της επιστολής της 11ης Μαΐου. Η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι ικανοποιημένη όσον αφορά κάποιες απαντήσεις που πήρε σε εκείνο τον τριμερή διάλογο, εκείνη τη σκοτεινή νύχτα που λέγατε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σεβάστηκε ορισμένα πράγματα που είχαν συζητηθεί τότε. Η πολιτική συμφωνία δεν αντικατοπτρίζεται δηλαδή, πιστεύω τελικά. Οπότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να το διορθώσει αυτό. Αυτά είναι τα σημεία που είχα να αναφέρω και υπάρχουν και κάποια άλλα που έχουν να κάνουν με την ουσία της δικιάς μου της ερώτησης. Ευχαριστούμε Κάθριν. Ο κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Κομισιόν και της ΑΕΟΠΑ, ιδίως για τα φιλικά λόγια του Μάριο Νάβα, ότι υπήρξε ο ήρωας τη νύχτας εκείνης βρίσκω πολύ ε, ευγενική την παρατηρησή του. Τώρα για το θέμα της ισοδυναμίας τρίτων χωρών. Να θέσω ορισμένα θέματα. Ήδη κατ' επανάληψη έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταχεία υποβολή των σχεδίων στη βάση των διαφόρων νομοθετικών πράξεων και είναι και σημαντικό για μένα να μην σημειωθούν άλλες καθυστερήσεις διότι το καθεστώς Solvency 2 πρέπει να μπορεί να είναι στην αφετηρία, να αρχίσει να ισχύει δηλαδή από 1η Πρώτου 2016. Πρέπει λοιπόν να προωθηθούν οι προσπάθειες διότι η ασφάλεια σχεδιασμού είναι το κυριότερο στοιχείο. Η κυρία ε, Στάιλερ τα εξήγησε και βεβαίως ενδιαφέρει αυτό και την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Βιομηχανία, τον Ευρωπαϊκό Ασφαλιστικό Κλάδο. Το σχέδιο της ΑΙΟΠΑ υπάρχει ήδη υπόψη της Κομισιόν. Γι' αυτό και παρακαλώ την Κομισιόν να κάνει μια πρόβλεψη ήδη σήμερα από τις αποφάσεις λοιπόν για τις τρίτες χώρες τι μπορεί να αναμένουμε. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε μόνο μένα τις ισοδυναμίες τρίτων χωρών. Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών αφορά ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει λοιπόν να ακολουθούν τις εξελίξεις FSP και IIS. Στην περίπτωση των ΗΠΑ συνδέονται και οι συζητήσεις για μια λεγόμενη covered agreement, μια διεθνή συμφωνία. Λοιπόν, θα ήθελα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσω πού βρίσκεται και εάν προβλέπεται συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ashley Φόξ ε, της ομάδας ε, συντηρητικών και ε, δημοκρατών, ECR. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προχώρησε ταχύτερα στις πράξεις για τις οδυναμίες τρίτων χωρών, γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείε έχουν ε, δουλειές και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση και χρειάζονται τι προφορίες αυτέ το δυνατόν συντομότερο. Παρακαλώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει ταχύτατα. Δεύτερο, Υποστηρίζω τις προσπάθειες που γίνονται για τον υπολογισμό του κινδύνου των μακροπρόθεσμων επενδύσεων των επενδυτικών ταμείων. Με ανησυχεί τρίτον τα έγγραφο της ΑΙΟΠΑ που προβλέπει αξίες spread πολύ υψηλότερες από αυτές που πρότεινε στον τριμερή διάλογο Omnibus 2 η ΑΙΟΠΑ και που έχουν δημοσιευθεί ήδη από το Μάιο 2014. Πολλές αξίες έχουν αυξηθεί κατά πάνω από 30% λόγω της πρόσφατης αυτής προσέγγισης και τα σπρέντα αυτά μειώνουν την προσαρμογή και επομένως τη συμφωνία που καταλήξαμε προηγούμενα. Γιατί λοιπόν προβλέπει τώρα με τόσο μεγάλη σημαντική αύξηση τα θεμελιώδη spread σε σύγκριση με αυτά που πρόβλεπε στην αρχική της ε, εκτίμηση και συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι στην συμπράξεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί υπό την ε, Solvens 2. Για την ώρα βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο θέμα, Άσλη, Τη ισοδυναμίας. κοιτάξτε, έκανα τι ερωτήσει τώρα για να μην ξαναπάρω το λόγο μετά. Νιουενχάιζεν των Φιλελευθέρων. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ε, ε, εκφέρατε το όνομά μου. Ερώτηση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιωτικά ταμεία. Δύο μέρη θα έχει ερώτησή μου. Πρώτο, όπως διαλαμβάνεται και στο πράσινο ε, έγγραφο, στο πράσινο βιβλίο, και η θεσμική επενδυτές με μακροπρόθεσμα holding, αλλά υπάρχουν και ορισμένες ρυθμιστικοί, ορισμένοι ρυθμιστικοί περιορισμοί που μειώνουν οι προβλέψεις για κεφαλαϊκές απαιτήσεις που προβλέπει η οδηγία Solvency 2 αποτελούν φραγμό για τις επενδύσεις ασφαλιστικών εταιρείων. εταιριών Μπορεί όμως να αποθαρρυνθούν τα συνταξιωτικά ταμεία από το να επενδύσουν σε relatives, αλλά ο Διονύος δεν είναι καθόλου σίγουρος ότι έχει ακούσει καλά. Και θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κατεξιότητες πράξεις. Και δεύτερο ερώτημα, ευρύτερο τώρα, χρειάζεται να δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς θα προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ενισχύσει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρώπη. Δεν βλέπω την κυρία Ματίας βέβαια της ομάδας ε, της Νοτικής Αριστεράς. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Σβέν Γκίγκολτ των Πρασίνων. Μια διευκρίνηση. Τώρα συζητάμε τα τρία θέματα μαζί ή το καθένα χώρια. Γιατί λίγο έχασα το σειρά. Το πρώτο, το πρώτο μόνο. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα, μάλιστα. Είχα μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Μπορείτε να μας πείτε, δώσετε τον πλήρη κατάλογο για το ποιες άλλες χώρες σχεδιάζουν ε, κανόνες αντιστοιχίας, ε, πού, έχουν, πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για παράδειγμα με την Κίνα. Μπορείτε να μας πείτε. Δεύτερον, Θα ήθελα να πω ότι ένα θέμα που πιστεύω ότι ίσως επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε, επειδή βλέπω και τον Μιχαήλ Τόιρερ εδώ, ε, στο πλαίσιο της Επιτροπής Τάξη, υπάρχει φυσικά κάποια σχέση ανάμεσα στην ρυθμιστική συνοχή και από την άλλη πλευρά κάποια αρχές επιθετικής φοροαποφυγής. Είδαμε κάποιες πρακτικές τέτοιες στις χώρες ενώ άλλες χώρες ήταν πολύ επιτυχείς και συνέδεσαν διάφορα θέματα για να βρουν κάποιες συμβιβαστικές στο επίπεδο της φορολογίας. Αύριο το πρωί η Ελβετία θα ε, υπογράψει την Συμφωνία ανταλλαγή Πληροφοριών με την Ένωση και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτό ποτέ δεν θα είχε συμβεί αν οι ΙΠΑ δεν ήταν έτοιμες να ασκήσουν πολύ μεγαλύτερη πίεση σε άλλους τομείς. Για τον τομέα λοιπόν των ασφαλίσεων η Επιτροπή η Τάξη θα πρέπει να εξετάσει κάποιες πρακτικές ε, επιθετικής φοροαποφύγης. Μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει, αλλά είναι ένα από τα δυνητικά παρόμοια μέτρα και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε, αν και κατανοώ ότι δεν είναι αυτή η εντολή της Επιτροπής και άρα δεν αναμένω να το σχολιάσετε. Νομίζω ωστόσο πως είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Δεν θα το σχολιάσω, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις για τις δυνατότητες των ΙΠΑ και κατά πόσο αυτά ταιριάζουν με την Ένωση. Ποιος είναι επόμενος, ο Μάριο. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω με τη σειρά που τέθησαν οι ερωτήσεις. Κυρία Στήλερ, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Βεβαίως, νομίζω πως έχω σημειώσει πολύ καλά τις ανησυχίες σας και τις ανησυχίες των συναδέλφων σας, ε, δηλαδή χρόνος και δέσμη. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν προσεχώς, το, το προσεχώς σημαίνει ότι ακριβώς ε, σύντομα θα ληφθούν. Πάντως, δεν θέλω να σας πω αν είναι μέρες ή εβδομάδες, πάντως σίγουρα δεν θα είναι μήνες. Οι επικείμενες λοιπόν αποφάσεις αποδεσμεύονται αναείδος αντιστοίχησης. Είναι σαφές δηλαδή ότι έχουμε από τη μια πλευρά μια νομική πράξη για πλήρη αντιστοίχηση και από την άλλη πλευρά έχουμε τη νομική πράξη για ε, για προσωρινή αντιστοίχηση. Και αυτό σέβεται νομίζω το πνεύμα αυτής της συμφωνίας που ήταν σκοτεινό μόνο επειδή ήταν Νοέμβριος μήνας αλλά όχι τον, λόγω των όσων συνέβησαν εντός αιθούσης όπου βρήκαμε μια πεφωτισμένη ισορροπία. Για το μέλλον τώρα τη μελλοντική πράξη που προβλέπεται για το φινόπορο μπορώ να επαναλάβω μόνο την ε, προτίμησή μας να είναι ακόμα πιο αποδεσμευμένες ε, αναχώρα. Ο κύριος Μπάλτς και ο κύριος Γκίκολτ με ρώτησαν αν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένος για τις χώρες. Αυτή τη φάση όχι, διότι αυτή, τώρα το εξετάζουμε και δεν έχουμε απόλυτα ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά σίγουρα Από τότε στον κύριο Μπάλτσε θα ξανασυναντηθούμε, συναντιόμαστε κάθε μήνα και ε, δεν παραμελώ να έρχομαι γιατί βρίσκω ότι είναι πολύ βοηθητικό για μας την Επιτροπή. Αλλά και ως πολίτης το βρίσκω πολύ θετικό, πολύ βοηθητικό ε, γιατί πρέπει όντως να σας ενημερώνουμε ε, μόλις θα έχουμε πιο νέες πληροφορίες από την ΑΙΟΠΑ πράγμα που το οποίο έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο. Έχουμε τουλάχιστον δύο-τρεις ακόμα δηλαδή συναντήσεις πριν να ε, ολοκληρωθεί. Και σίγουρα δεν θέλω να υπάρξουν εκπλήξεις. Όπως σήμερα ξέρετε τι θα συμβεί. Όπως σας είπα είναι θέμα μερών ή εβδομάδων το πολύ, αλλά γνωρίζετε ακριβώς τι θα γίνει. Τι είδους ισοδυναμία ή αντιστοιχεία, για ποιες χώρες, ε, κύριε Φόξ, συμμερίζομαι την απογοήτευσή σας για την καθυστέρηση και εγώ θα ήθελα πολύ αυτή η καθυστέρηση να μην είχε συμβεί, όμως συνέβη και ε, σας παρακαλώ να με πιστέψετε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελεγχιστοποιήσουμε τις καθυστερήσεις και να ε, με την άδειά σας θα ήθελα να απαντήσω σε εσά και στην κυρία Φανίεν Χόιζεν. Θα σας απαντήσω αργότερα το θα μιλήσουμε για την LTIF. Ωραία. Θέλετε κάποιος να προσθέσει κάτι για το πρώτο θέμα, την ισοδυναμία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω έχει να κάνει με την καθυστέρηση που ανεφέρθη. Η ΟΠΑ εξέδωσε πρόσφατα γνωμοδότηση για τα ιστορικά πρότυπα, μοντέλα και προέβησε συστάσεις όσον αφορά τους χρήστες των εσωτερικών μοντόλων που θα μπορούσαν να προβούν σε υποθέσεις για τις κατεξοδότητες συμπράξεις όταν αυτές έχουν εκδοθεί και σε σχέση με την ισοδυναμία στο πλαίσιο αυτό. Είναι ένα τεχνικό, μια τεχνική φύση παρατήρηση, αλλά το γνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε λοιπόν στην κατεξοδότηση πράξη σε σχέση με τα LTIF. Ε, που τροποποιεί την, την, την ε, απόφαση για το Insolvency 2. Κατανοούμε ότι η Κομισιόν σκοπεύει να ε, τροποποιήσει τον σχετικό κανονισμό πριν το καλοκαίρι του 2015 με στόχο να, να ενσωματώσει τον πρόσφατα μεταρρυθμισμένο κανονισμό για το Ταμείο Φερεγγιότητας που θα ενσωματωθεί στο Insolvency 2 και θα έχουμε συγκεκριμένο ε, ε, κίνδυνο που θα αναλαμβάνουν οι ασφαλιστές Έχουμε δηλαδή τους κανονισμούς 145 του 2014 και 346 του 2013 που θα ε, ενσωματωθούν στο Insolvency 2 κατανοούμε ότι τα κράτη-μέλη μέχρι στιγμής δεν είχαν αντίρρηση γιατί η ΑΙΟΠΑ δεν ερωτήθηκε από πλευρά τη Κομισιόν για input. Οπότε ξεκινάμε από την Κομισιόν. Μάριο, μπορείς να μας κάνεις μια σύντομη επισκόπηση. Ναι, να σας πω ότι θέλουμε εδώ να ενεργήσουμε για αυτό το θέμα και όπως είπατε Πρόεδρε, η ΕΛΤΙΦ, ε, το Ευρωπαϊκό Μακροπρόθεσμο Επενδυτικό Κεφάλαιο δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί. Αν υπήρχε, όταν τα είχαμε διαπραγματευτεί αυτά, δεν θα ήμασταν εδώ να τα συζητάμε, γιατί εξ αρχής τα είχαμε προτείνει και μάλλον θα έχει γίνει και δεκτό από όλους τους μπλεκόμενους από την αρχή, αμπινίτσιο, θα είχαμε προτείνει λοιπόν την ίδια μεταχείριση όπως το κεφάλαιο κινδύνου και το κεφάλαιο, ε, το κοινωνικό κεφάλαιο. Ε, δυστυχώς δεν υπήρχε τότε, αλλά αυτό ευτυχώς μπορούμε να το διορθώσουμε αρκετά εύκολα με μια τροποποίηση μια τροπολογία. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να το δούμε και έρχομαι άμεσα στο ερώτημα του Κόνρατ, ότι δηλαδή θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο της ε, στάθμισης. Ε, να βρούμε δηλαδή τη σωστή στάθμηση, ε, για, έτσι ώστε να μπορούν να επενδύουν τα δημοσιονομικά θεσμικά όργανα. Έχουμε εδώ δηλαδή μια ευκαιρία που είναι η δυνατότητα ενός ασφαλιστή να αναλάβει πιο μακροπρόθεσμους κινδύνους από ότι άλλοι εταίροι ή άλλη θεσμοί. Και αυτές οι δυνατότητες, αυτές οι ευκαιρίες θα πρέπει να ε, μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε το LTIF. Αλλά επίσης, αυτό που ζητήσαμε από την ΕΙΟΠΑ, όπως είχα την ευκαιρία να σας αναφέρω, είναι ότι ζητήσαμε τη συμβουλή τους για το ποιες είναι οι απόψεις τους όσον αφορά τους ασφαλιστικούς επενδυτές στα προγράμματα υποδομής, στα, στα project υποδομής. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια οικονομική πράξη, αλλά δεν πρόκειται για απομονωμένη πράξη. Εντάσσεται στην ανάγκη στάθμισης των κανονισμών ώστε να καλύπτουν τους απαραίτητους μακροπρόθεσμους, τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που μπορούν να κάνουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να τους κάνουν. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει κάτι να προσθέσει. Η ΑΙΟΠΑ καλωσορίζει την ε, πρωτοβουλία αυτή για την εξέβρεση μακροπρόθεσμων λύσεων για τους ε, επενδυτές αυτούς. Ε, για την ΑΙΟΠΑ είναι σημαντικό αυτή η πρωτοβουλία να εξασφαλίζει ότι τα, η χρέωση του κινδύνου να είναι αντίστοιχη με τον πραγματικό κίνδυνο. Καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο όχημα όπως το ΕΛΤΙΦ θέλει να στηρίξει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τις υποδομ, επενδύσεις σε υποδομές ώστε να υπάρχει έκθεση σε μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού. Να σας πω δύο λόγια για τις υποδομές εφόσον αναφέρθηκε από τον κύριο ε, Νέδερ και ήταν και θέμα το οποίο έθιξε η κυρία Νέιγενχάουζεν για την επέκταση δηλαδή των ρυθμίσεων αυτών. Η ΕΙΟΠΑ σήμερα δεν εστιάζεται μόνο στη στάθμιση του κεφαλαι... της κεφαλαϊκής χρώσης, πράγμα το οποίο εξαρτάται από τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί για πραγματικές επενδύσεις. Είναι σημαντικό οι ασφαλιστές να έχουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη ώστε να αποσωτικοποιήσουν και να χειριστούν τους κινδύνους. Όπως υπόθηκε ήδη, η ΕΙΟΠΑ εργάζεται ήδη συμβουλεύοντας την Επιτροπή για την Ανάπτυξη μιας ε, τάξεις ε, επενδυτικών ε, στοιχείων ενεργητικού στις υποδομές και έτσι ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια για τις επενδύσεις αυτού του τύπου. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι θα δώσω τη λόγο στην εισηγήτριά μας, την Κάθριν. Εάν εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι κάποιοι άλλοι έχουν πιο πολλές ανησυχίες και άρα ας χρησιμοποιήσουν ε, το χρόνο για να απαντηθούν ερωτήσεις. Κόρα, η ερώτησή σας ε, απαντήθηκε ο Μάικλ, αν και δεν είναι αυτός ο κανόνας. Τέλο πάντων, θέλω να δω οι άλλοι σκιώδη Άσλι. Ε, τότε ο Μάικλ. Catch the eye. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, Μπορείτε παρακαλώ σύμφωνα με τη στάθμιση κινδύνου να μας πείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις και μπορείτε να μας ενημερώσετε για τον τύπο της στάθμισης και αν ναι, πότε μπορείτε να το κάνετε αυτό. Πρόεδρος, δεν ζητάει κανένας άλλος το λόγο. Συνεπώς, Μάριο, μπορείς να απαντήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι αυτή η στάθμιση πρέπει να έχει πολύ γερή Θέλουμε λοιπόν να δούμε έναν δείκτη για τις τιμές των equities. Είναι ένα, τεχνική ερώτηση, τεχνική απάντηση θα πάρετε. Το LPX NAV 50. 50. Και η εμπειρική ανάλυση του δίκτυα αυτού για μια μεγαλύτερη περίοδο από το 2003 μέχρι το 2013, για 11 χρόνια δηλαδή, δείχνει ότι 99,5% είναι πολύ κοντά στο 39% αξίας στάθμισης που δίνουμε. Συνεπώς, η βάση, τα θεμέλια του ΕΛΤΙΦ συνάδει με τον κίνδυνο που αναφέρουμε. Σας είπα, 11 χρόνια ο δείκτης των ιδιωτικών equities, όλα έγιναν, είναι καλές χρονιές αυτές δηλαδή, έτσι. Οι πρώτες χρονιές ήταν καλές, οι επόμενες ήταν λιγότερο καλές και μετά Ξανά καλά. Έχουμε λοιπόν γέρη βάση και ευχαρίστως να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης συζητήσαμε σε πρόσφατη συνάντηση πριν από λίγους μήνες με τις χώρες μέλη και με το Κοινοβούλιο. Ο Ιβο Βανές ήταν εκεί από πλευράς της Γραμματείας ΕΚΟΝ. Οπότε έχουμε δώσει τις λεπτομέρειες πολύ ανοιχτά. Αλλά ευχαρίστω είμαι στη διάθεσή σας να τα επαναλάβω αν θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ Μάριο. Και συγγνώμη να προσθέσω κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φόξ για την θέση του που μας στηρίζει. Ο κύριος Ρέχει και εκείνο κάτι να προσθέσει. Ναι, δεν μας ζητήθηκε να εξετάσουμε το θέμα των relatives. Ωραία, ερχόμαστε στο τρίτο, Θερμοστικές πράξεις. Για δομές επιτοκίων ανευκινδύνου, διορθώσεις. Θα έπρεπε να αποφεύγεται τεχνητή ρευστότητα και να προσφέρει κίνητρα για καλή διαχείριση κινδύνου. Συνεπώς, το σημείο κίνησης για να καταλήξουμε στους αριθμούς όσον αφορά το ευρώ θα χρειάζεται 20 χρόνια ορίμανση. Ιδιαίτερα όσον αφορά το ευρώ θα πρέπει η σύγκληση να γίνεται με βάση 40 χρόνια ορίμανση και να μην υπάρχει διαφορά πάνω από τρεις μονάδες βάσης. Ελπίζω όλοι να καταλάβατε τι είπα, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα για άλλο νομίσματα εκτός ευρώ, το σημείο κίνησης και η σύγκληση μπορεί να είναι διαφορετική. Για το UFR Είμαστε στα 4,2%. Έχετε το λόγο. Αρχίζουμε τώρα με την ΙΟΠΑ. Και μετά θα πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά βέβαια ο εισηγητής, η εισηγήτρια μάλλον και σκιώδης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε, η νομοθεσία μας έχει αναθέσει να δημοσιεύουμε τεχνικές πληροφορίες όσον αφορά τους δείκτες βάσει της Solvency 2. Όσον αφορά τους κινδύνους, οι διορθώσεις στη ρευστότητα και οι υπολογισμοί πρέπει να είναι κατάλληλοι. Η οποία αποφάσισε να δημοσιεύει ήδη την τεχνική ε, πληροφορία και προετοιμάζουμε ό,τι περιλαμβάνεται στο Solvency 2, την ασφάλιση και την αντασφάλιση δηλαδή. Οι τεχνικές πληροφορίες που δημοσιεύουμε ε, θα είναι όταν θα έχει συμπεριληφθεί δημοσίευση της ίδιας της Επιτροπής στις εφαρμοστικές πράξεις. Αυτό θα αρχίσει από το 2016 και η δημοσίευση θα γίνεται κάθε τρεις μήνες. Η ΟΠΑ όμως θέλει κάθε μήνα να δημοσιεύει τα στοιχεία. Ο υπολογισμός τώρα που κάνουμε βασίζεται στους στόχους της ανταπόκρισης και της σταθερότητας. Το πρώτο σημαίνει ότι όλοι οι διαφερόμενοι ασφαλιστές και αντασφαλιστές μπορούν να αντιδράσουν στους υπολογισμούς. Γι' αυτό και δημοσιεύουμε τεχνική τεκμηρίωση με την μεθοδολογία μεταξύ άλλων. Και σταθερότητα σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε την ρευστότητα να την υπολογίσουμε χωρίς τα τεχνικά στοιχεία και μετά από διαβούλευση. Οι τεχνικές, τα τεχνικά στοιχεία τα εξετάζουν και οι ασφαλίσεις και τα ασφαλίσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν και αυτό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you very much. Mario for the Μάλιστα, τη Κομισιόν. Όπως είπε και ο κύριος Ρέι όχι προηγούμενη βραδιά, αλλά λίγο πριν, όταν είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό, κέριο θέμα βέβαια, το οποίο δίνει στην ΑΙΟΠΑ και μεγαλύτερες ευθύνες για τον υπολογισμό του, της αναλογίας αυτής, του rate αυτού και βεβαίως και διαφάνεια και ικανότητα των άλλων να μπορούν πρώτα να κατανοήσουν και δεύτερον να επαναλάβουν τον υπολογισμό, αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας. Πολύ χαίρομαι, όπως είπε ο κύριος Ρέι, ότι η ΑΕΟΠΑ υποστηρίζει την σταδιακή εφαρμογή της Solvency 2, δημοσιεύοντας ήδη τους συντελεστές αυτούς, που βεβαίως δεν είναι ακόμα δεσμευτικοί, δεν είναι ακόμα τμήμα της νομοθεσίας, ωστόσο έχουν δημοσιευτεί ήδη και δημοσιεύονται ανά μήνα Βέβαια η νομοθεσία λέει ένα τρίμηνο, πάντως αυτή δημοσιεύονται ήδη από ε, τώρα για κάθε μήνα και μας βάζει σε καλό δρόμο για την ε, θέση ισχύ της Solvency 2 από 1η Πρώτου 2016. Ευχαριστώ. Η Κάθριν Στίχλερ. Σχόλιο, ναι. Διαφάνεια, πολύ σημαντική. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, απλώς η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε βέβαια τις εκατεξουσιοδότηση πράξεις που τις συζητήσαμε αρχές Δεκεμβρίου εδώ για την Solvency 2 και μεταξύ αυτών και τα μέτρα για την δομή των επιτοκίων. Και γι' αυτό ευχαριστώ και την Κομισιόν και την ΑΕΟΠΑ που ξαναθέτουν το θέμα ακόμη και αν η πολιτική συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων είναι σαφής και δεν μπορεί να τροποποιηθεί με, απλούς, με απλές ε, εκτελεστικές πράξεις. Δεν αφήνω διάφορο τα θέματα αυτά βεβαίως κανένα ενδιαφερόμενο και επειδή η, ο ασφαλιστικός κλάδος ε, θέλει ε, προβλεψιμότητα. Θα πρέπει και η πορεία των επιτοκίων να είναι σαφείς, διότι είναι και οι προβλέψεις σημαντικές και κυρίως για το τέλος τους. Γνωρίζουμε πότε άρχισε η παρούσα φάση των ε, χαμηλών επιδοκίων και αυτό οφείλουμε να το θέσουμε υπόψη και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα έπρεπε να είχε προσφυθεί τότε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά βεβαίως ο πρόεδρος της κ. Ντράγκη γνωρίζει το θέμα ήδη από τους διάφορους νομισματικούς διαλόγους που έχουμε διαξαγάγει μαζί του και εδώ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Δεν κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο να τον προσκαλέσουμε τότε. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε βεβαίως ότι ο κύριος Δράγκη θα παρακολουθεί και τις συζητήσεις μας αυτές. Άσλι Φόξ δεν θέλει, οι φιλελεύθεροι δεν θέλουν, οι κομμουνιστές είναι απόντες. Α, Σβέν, εδώ είσαι πάλι των Πρασίνων, ο κ. Κίγκολ δηλαδή. Η συζήτηση αυτή και είπε και ο Μπούρκαρτ Μπάρτ σωστά ότι ήδη πετέλεσε θέμα στις νομοθετικές μας συζητήσεις αλλά παρόλα αυτά το πώς θα θεσπίσουμε τους ε, εναλλακτικούς συντελεστές και σε ποια βάση και γιατί άραγε βάζετε 4,2% αυτό είναι άλλη υπόθεση. Δεν θεσπίσαμε το επίπεδο και καλό είναι που ο νομοθέτης δεν πιστεύει ότι γνωρίζει ποιος είναι ο τελικός συντελεστής. Αυτό που είναι ωστόσο εκπληκτικό, εάν συγκρίνετε τον πίνακα που σας δείχνω τώρα που, ε, εδώ στο έγγραφο με την καμπύλη των επιτοκίων και το ultimate forward rate και το ρυθμιστικό συντελεστή που εφαρμόζεται τώρα στις ευρωπαϊκές ε, ασφαλίσεις θα δείτε μια μεγάλη διαφορά και η μεγάλη διαφορά αυτή σημαίνει ότι η αγορά πιστεύει κατά βάση ότι δεν είναι βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που συμπιέζουν τα επιτόκια, αλλά ότι είναι μια εξέλιξη διαρκής που θα παραμείνει. Και αυτό σημαίνει ότι η ΑΙΟΠΑ πιστεύει ότι γνωρίζει καλύτερα το μέλλον των αγορών από τις ίδιες αγορές. Από αυτά που πιστεύουν οι αγορές ότι τις αναμένει στο μέλλον. Αυτό χρειάζεται όμως αιτιολόγηση διότι οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν και την αρχή της ε, επιμέλειας. Γι' αυτό και θέλω να ακούσω από την ΑΕΟΠΑ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αιτιολογούν αυτή τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των, ε, των συντηρηστών της αγοράς και των προσδοκιών τους και του δικού της Ultimate Forward Rate και αυτό είναι σημαντικό βέβαια και για τον εισηγητή. Διότι εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες, αν τους ζητηθεί δηλαδή, να μην έχουν επαρκείς προβλέψεις, αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ε, ε τις μελλοντικές αποδόσεις τους καθώς και το μέλλον της οικονομίας. Και γι' αυτό ρωτώ, με ποιον τρόπο κατέληξε η ΟΠΑ στο 4,2% και αν το 4,2% αποτελεί πράγματι το προϊόν επιμέλειας ή απλά συζητήσεων στο Εποπτικό Συμβούλιο που δεν ήθελε να εκδώσει άσχημα νέα. Τέλος, με ανησυχούν ε, ακόμη ορισμένες από τις διαφορές μεταξύ των swap rates και των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων που στη βάση τους υπολογίζονται τα rates. Και εδώ η προσαρμογή του credit risk για κρατικά ομόλογα της Ουγγαρίας είναι μόνο σε 10 ποσοστιαίες μονάδες. Ενώ το rating της Ουγγαρίας είναι διπλό β. Και η αξιολόγηση της Βραζιλίας που είναι τριπλό β, εκεί το κρατικό ομόλογο, το credit risk adjustment, είναι 35% μονάδες βάσης. Το θεωρείτε λοιπόν δικαιολογημένο αυτό και το θεωρείτε ότι είναι προϊόν της άσκησης της ορθής επιμέλειας. Να επανέλθει η ΟΠΑ λοιπόν και να μας εξηγήσει πώς κατέληξαν σε αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία για μένα αποτελούν ένιγμα αφού πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αγορέ και όχι να πιστεύει ότι τα κράτη γνωρίζουν τις, ε, τους κινδύνους καλύτερα από τις αγορές. Δεν έχω αλλού λέει ο πρόεδρος, που να ζητούν το λόγο, γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον Justin Day της ΑΙΟΠΑ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ γιατί ε, όντως πρέπει να απαντήσω σε διάφορες ερωτήσεις. Πριν στραφώ στραφόμαστε αυτό, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να απαντήσω στα όσα είπε ο κύριος Φόκ την πρώτη του παρέμβαση, ότι μίλησε για το επίπεδο του βασικού spread. Ε, να εξηγήσω ποια είναι η βάση για τις αλλαγές στα νούμερα. Το 2013 η ΟΙΟΠΑ εκπώνησε την έκθεσή της για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και τη συμβουλή της ΑΙΟΠΑ βέβαια που ε, προηγήθηκαν τις απόφασες Omnibus 2 που τώρα ορίζει τι απαιτείται για τις μακροπρόθεσμες εγγύησεις και βασιζόμαστε στην μεθοδολογία που σχεδίασαν οι συνομοθέτες όπως αυτή εκφράζεται στο μήνυμα 2. Ναι, τα νούμερα είναι λοιπόν διαφορετικά αλλά αντικατοπτρίζουν την μεθοδολογία, την επιθυμητή μάλλον μεθοδολογία. Έπειτα, όσον αφορά τα ερωτήματα του κύριου Κίγκολντ, θα προσπαθήσω να απαντήσω Καταρχήν θέλω να εξηγήσω πώς ε, ε, προκύπτει το ultimate forward rate ε, έπειτα κατά πόσο λαμβάνουμε υπόψη τα χαμηλά επιτόκια και ποια είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε. Το συγκεκριμένο ερώτημα για το πίνακα και για την προσαρμογή του πιστοτικού κινδύνου για την Ουγγαρία. και το κατά πόσο το ποσοστό θα είναι 4,2 ε, που είναι ψηλότερο ε, προέκυψε. Αυτό γίνεται με βάση την Solvency 2 και τις συμπληρωματικές εφαρμοστικές πράξεις που θα ακολουθήσουν. Οι κατεξιδότητες συμπράξεις απαιτούν να ε, το μοιράσουμε αυτό ως το σύνολο του αναμενόμενου μακροπρόθεσμου ε, ε, επιτοκίου και αυτό σχετίζεται με το στόχο πληθωρισμού της ΕΚΤ, δηλαδή 2% και τώρα ξέρουμε ότι καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούν σε αυτό το στόχο. Μα, τώρα ο το μακροπρόθεσμο επιτόκιο, πραγματικό επιτόκιο είναι 2,2% και η τεχνική τεκμηρίωση σημειώνει ότι η μέση πραγματική απόδοση στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα ήταν 3,2% για διάφορες χώρες. Έχουμε δηλαδή ε, βασιστεί σε αυτά τα στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Ultimate Forward Rate 4,2% χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια του εκπόνησης του Omnibus 2. Τώρα, για τις παρατηρήσεις σας ε, που αφορούν τα ισχύοντα χαμηλά επιτόκια. Εμείς ε, δεν υποστηρίζουμε ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα, απλά εμείς εφαρμόζουμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό όλων αυτών. Σύμφωνα με την κατεξοδότηση πράξη θα πρέπει ε, αυτά τα επιτόκια να είναι σταθερά και να αλλάζουν με βάση τις ε, αλλαγές της μακροπρόθεσμες της προσδοκίας και πάλι πρόκειται για το άρθρο 47. Και όταν η κατεξοδότηση πράξη αναφέρεται στα μακροπρόθεσμα επιτόκια, αναφέρεται σε, διάφο... σε αρκετές δεκαετίες όσον αφορά το ασφαλιστικό παθητικό Μιλάμε για 60 χρόνια ε, προοπτική και αυτό είπα προηγουμένως ότι δηλαδή ο αντίκτυπος του UFR 4,2% του Ultimate Forward Rate δεν ε, αφορά τις, ε, μάλλον δεν αφήνει απ' έξω τις πρώιμες την πρώιμη ορίμανση ή ε, λήξη ασφαλιστικών συμβολέων, αλλά υπολογίζει με βάση μια προοπτική αρκετών δεκαετιών. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι αυτό το επιτόκιο είναι συνέπεια για, μάλλον θα έχουν συνέπειες όσον αφορά τις, ε, την, τη, τη, λήξη των συμβολέων σε αρκετές δεκαετίες και όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες, η αναμονή, οι, ε, προεκβολές που μπορεί να έχουμε. Πρόσφατα, μάλλον υπάρχει ένας ε, χάρτης ε, που κυκλοφορεί και υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια που προβλέπονται. Να σας πω ότι ένας από τους στόχους Τη δική μας προσέγγιση είναι η δυνατότητα επανάληψης, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε μια ειδική εμπειρογνωμοσύνη και κρίση, ώστε να μπορούν τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη να, να επαναλάβουν και να αντιγράψουν αυτά τα ποσοστά. Στην κατεξοδότηση πράξη και σε άλλες νομοθεσίες μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα επιτόκια ε, μέχρι πριν 20 χρόνια τα, τελευταία, τον τα επιτόκια των τελευταίων 20 ετών. Αυτά ορίζονται μέσα στη μεθοδολογία που μόλις σας περιέγραψα και γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε προβολές με βάση τα στοιχεία των τελευταίων 20 ετών. τελευταία σας παρατήρηση αφορούσε την, την προσαρμογή για την Ουγγαρία και την προσαρμογή του πιστατικού κινδύνου για την Ουγγαρία. Και πάλι η κατεξοδότηση πράξη απαιτεί τον ορισμό ε, του πιστοτικού κινδύνου με, εντός κάποιων παραμέτρων. Και στην περίπτωση της Ουγγαρίας εμείς λάβαμε την, το πιστοτικό κίνδυνο για το ευρώ και το εφαρμόσαμε στους, ε, στη χαμηλότερη δυνατή κλίμακα, δηλαδή στους, ε, στις 10 μονάδες βάσης. Έτσι υπολογίσαμε το πιστοτικό κίνδυνο για την Ουγγαρία και ευχαριστώ Πρόεδρε, εδώ ολοκλήρωσα την απάντησή μου. Ευχαριστώ, η Κομισιόν θέλει να προσθέσει κάτι, όχι. Εγώ μπορώ να επανέλθω όμως στην ερώτησή μου. Μα ακούσατε μόλις μία μακρά απάντηση. Όχι, η απάντηση που δεν απαντήθηκε κατά πόσο είστε έτοιμος να επανεξετάσετε τη μεθοδολογία σας για να αποφύγετε την εντύπωση που δίνετε ότι απλά είστε μια απλή, ένας απλός οργανισμός ε, υπολογισμού των επιτοκίων. Τα επιτόκια όμως, το αποτέλεσμά σας μάλλον, είναι πολύ μακριά από τις προσδοκίες και την προβολή των αγορών. Μήπως λοιπόν πρέπει να αναθεωρηθεί η μεθοδολογία σας. Μήπως σκεφτείτε να αλλάξετε τη μεθοδολογία σας. Σύντομη απάντηση. Εγώ το μήνυμα που πήρα ήταν ότι έπρεπε να μου περιγράψετε τη μεθοδολογία. Εν πάση περιπτώσει. Ίσως εγώ να μην κατάλαβα καλά. Ο κύριος Ρέι. Θα ήθελα να σας πω ότι, ναι, εξηγώ πώς φτάνουμε στο 4,2 UFR, προθεσμιακή ισοτιμία, ultimate forward rate. Αυτό πρέπει να ορίζεται για να εξασφαλιστεί το για να υπολογιστεί η ασφάλεια των προβολών και των υπολογισμών. Εμείς ορίζουμε ε, μάλλον έχουμε και τηρούμε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό δεν απαιτεί αλλαγή στο UFR. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να σας δώσω για το θέμα της μεθοδολογίας, κύριε Γκίγκολτ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίμαν και κύριε Ρέι. Εδώ θα διακόψουμε για λίγα λεπτά μέχρι ότου να ε, επανέλθει στην αίθουσα η διαπραγματευτική μας ομάδα από την ΕΦΣΥ. Thank you. So we are now going. Τώρα, λέει ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, θα προχωρήσουμε στο υπαριθμόν 5 τη ημερησίας διατάξεως που προβλέπει βεβαίω ένα ε, ιδιαίτερα σημαντικό θέμα Είναι λοιπόν όπως έλεγα πολύ ε, σημαντικό και βεβαίως υποτίθεται ότι θα ψηφίσουμε. Η κυρία Περέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να μου επιτρέψετε να ζητήσω από τους συναδέλφους των άλλων πολιτικών ομάδων να δεχθούν αναβολή της ψηφοφορίας για το σημαντικό αυτό θέμα. CRD3, CRD4, SSM, SRM και όλα τα σχετικά αρχικά τα οποία έχουμε συζητήσει καταλήξαμε να έχουμε σημαντική πλειοψηφία που απαιτέλεσε τιμή για την Επιτροπή μας καθώς και για το Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα υπάρχει κίνδυνος να σπάσουμε σε δύο μισά με πολύ περιορισμένη πλειοψηφία εάν ψηφίσουμε σήμερα όπως προβλέπετε. Σας παρακαλώ λοιπόν να δεθείτε, να ζητήσετε από το Λαϊκό Κόμμα, από τους Φιλελευθέρους και από τα άλλα πολιτικά κόμματα με τα οποία συμφωνούμε, να αναβάλουμε για μια εβδομάδα. Δεν θα προκαλέσει κανένα μείζον πρόβλημα όσον αφορά την ε, ημερολογιακή πορεία, το χρονοδιάγραμμα δηλαδή της νομοθεσίας και θα δώσει μια δυνατότητα να επιτευχθεί μια ευρύτερη πλειοψηφία στην στιγμή της ψηφοφορίας. Το έχω ζητήσει και διμερός, το ζητώ και δημοσία τώρα γιατί θα είναι και προς όφελος της Επιτροπής Οικονομικών αλλά και προς όφελος της ποιότητας των εργασιών του Ευρωκοινοβουλίου. Αν μπορέσουμε να αναβάλουμε σήμερα και να ψηφίσουμε σε μια εβδομάδα. Αυτά ήταν σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Ευχαριστώ κυρία Περέιρα. Αντιλαμβάνομαι το νόημα των λόγων σας όσον αφορά την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να επιτυγχάνουμε τις ευρύτερες δυνατές πλειοψηφίες ώστε να ενισχύεται η θέση μας μέσα στους τριμερείς διαλόγους. Βεβαίως την απόφαση για την αναβολή θα την λάβει ε, κυρίαρχα η Επιτροπή. Βεβαίως οι συντονιστές θα θέλουν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Μπάλτς για το Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην υπόθεση αυτή, όπως είπε και η Ελίζα Περέρα, έχω διεξαγάγει συνομιλίες και με την ίδια και με εσάς, Εξ ονόματος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, έχω να πω ότι προτιμούμε να ψηφίσουμε σήμερα, διότι θεωρούμε ότι το θέμα είναι πλέον όριμο για ψήφιση. Έχουμε διεξαγάγει άνω των 20 συναντήσεων μεταξύ των συντονιστών, σκεδών συγκριτών κλπ δεν κατορθώσαμε να φτάσουμε σε συμβασμούς και επομένως πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και πρέπει εν τέλει η Οικονομική Επιτροπή να μπορέσει να κρίνει για αυτό το σημαντικό όπως είπατε και εσείς και γι' αυτό εμείς επιθυμούμε να εμείνουμε στην σημερινή ψηφοφόρια. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Αντιλαμβάνομαι ποια είναι η θέση που αναπτύξατε. Αν Α, ο κύριος Λάμπερτς των Πρασίνων. Αν δεν υπάρξει ευρεία πλειοψηφία, υπάρχει η πιθανότητα να αποσύρει την πρότασή της. Θυμίζω την επιστολή Hill προς Timmermans η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν κολλήσει ο φάκελος λοιπόν αυτός, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιό της. Εγώ θα υποστήριζα το αίτημα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Βεβαίως διατηρώ τις επιφυλάξεις μου εάν μια εβδομάδα ακόμη θα μας επιτρέψει να καλύψουμε πολύ μεγάλα κενά μεταξύ εκείνων εξημών που πιστεύουν ότι χρειάζεται κάτι το σοβαρό επί του CRD και BRD. Αν όμως υπάρχει ε, περίπτωση να διεξαχθεί και άλλος διάλογος, εγώ βεβαίως είμαι υπέρ. Εγώ υποστηρίζω, η ομιλητρία, ε, τον ε, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και εξ όσων γνωρίζω από το κεφάλαιο, από, τον φάκελο αυτό, θεωρώ ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ψηφοφορία τώρα. Δεν θα υπάρξει συνένεση μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Συμπαρατάσσομαι λοιπόν με το ε, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η Γκουλάρ. Και εμείς είμαστε υπέρ της ε, ψηφοφορίας, διότι έχουν διεξαχθεί ε, μακρότατες συζητήσεις σε πνεύμα βεβαίω συμβασμού, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τάμουμε. Α, ο εισηγητής, ο κ. Χόκμαρτ του Λαϊκού Κόμματος. Κύριε Πρόεδρε, παρά τις μεγάλες διαφορές, δεξήχθηκαν πολλές επικοδομητικές συζητήσεις σε καλό κλίμα στην ομάδα διαπραγματεύσεων. Ξεκινήσαμε από μακριά και σε πολλά τμήματα της νομοθεσίας έχουμε προσεγγίσει οι μεν δε. Όπως είπε ο κ. Λάμπερτς προηγουμένως, είναι δύσκολο να πιθανολογήσω κι εγώ ότι θα επιτύχουμε να ξεπεράσουμε κάποιες γραμμές ε, διαχωριστικές που δεν καταφέραμε μέσα σε τόσες ε, μέρες και σε τόσες πολλές ε, συναντήσεις. Όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της ε, Οικονομικής Επιτροπής θα διασφαλίσουμε μια όθηση και μια νέα φορά στις ε, συζητήσεις με το Συμβούλιο. Αυτό που χρειάζεται είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε απόφαση. Έχει σημασία να διατηρήσουμε μια θέση υπεροχής απέναντι στο Συμβουλίο και εμείς να υπαγορεύουμε την ημερήσια διάταξη για να διατηρήσουμε έτσι τη δυνατότητα υπέρ των Ευρωπαϊκών Τραπεζών να συνεχίσουν να επενδύουν. Ευχαριστώ. Της Ενωτικής Αριστεράς. Είναι πολύ σοβαρά τα επιχειρήματα του Φίλιπ Λάμπερτ ότι μπορεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκαταλείψει την πρότασή τη, Επειδή όμω υπάρχει μέγα κενό μεταξύ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και των άλλων πολιτικών ομάδων που δεν είναι βέβαια ουσιώδη για να λυθούν τα προβλήματα του too big to fail βλέπω λοιπόν ότι είναι μεγάλο το κενό, μεγάλη απόσταση Δεν έχουμε εμεί καμία ιδιαίτερη προτίμηση. Εν τέλει λοιπόν, αν καταστεί αναγκαίο, προτιμούμε και εμείς να ψηφίσουμε σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Τζάνι. Σας ευχαριστώ. Έχουμε δουλέψει πολύ. Έχουμε κάνει σε συσκέψεις για να προσπαθήσουμε να ε, φέρουμε πιο κοντά τις απόψεις των διαφόρων ομάδων. Δεν είναι αυτό δυνατό και δεν πιστεύω πως μια παραπάνω εβδομάδα θα μας ε, είναι αρκετός χρόνος ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το παραπανήσιο βήμα για να μπορέσουμε ακόμη περισσότερο να φτάσουμε σε μεγαλύτερη πλειοψηφία και εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο να ψηφίσουμε σήμερα. Συμφωνώ με τον Φίλιπ ότι αν αυτό το σημερινό κείμενο δεν περάσει, υπάρχει ο κίνδυνος ε, η Κομισιόν ανάλογα με το πρόγραμμά της να το αποσύρει. Η ε, προσωπική μου άποψη είναι ότι να έχουμε ένα κείμενο ε, το οποίο έχει αποσυρθεί ή έχει εγκριθεί με τη θέση της, του εισηγητή ε, για μένα δεν έχει μεγάλη διαφορά, οπότε θα ήμουν υπέρ του να ψηφίσουμε τώρα. Εγώ βλέπω λοιπόν τότε ότι οι περισσότεροι θέλετε να ψηφίσουμε σήμερα. Αλλά αν θέλετε, αν οι σοσιαλιστές το ζητήσουν, μπορούμε να ψηφίσουμε πάνω σε αυτό το αίτημα. Ακόμα και αν εγώ βλέπω ότι υπάρχει πλειοψηφία, υπέρ του να ψηφίσουμε, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία ή θέλετε να ζητήσετε ψηφοφορία για την αναβολή. Ωραία, λοιπόν, να ψηφίσουμε κανονικά. Αναπροτείνω να κάνουμε πρώτα μια δοκιμή, να δούμε αν λειτουργούν όλα τα μηχανήματα. Βάλτε τις κάρτες σας στα μηχανήματα και κάνουμε δοκιμαστική ψηφοφορία. Έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚΑ. Ποτέ δεν είναι πολύ η, έλκα. η ΕΛΚ. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εντάξει λοιπόν, 40 ψήφοι. Ωραία, να βάλουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Όχι, όχι, αστιάκι, αστιάκι. Ναι. Ε, για να χαλαρώσουμε λίγο, είπα και εγώ ένα αστιάκι. Λοιπόν, και τώρα περνάμε στην πραγματική ψηφοφορία και ψηφίζουμε για τη συμβιβαστική α. Ποιοι είναι πέρ? Κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικός, άρχεται η ψηφοφορία. Okay, one is not voting, but okay, we can close the vote now. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίζουμε. So this clause Is rejected. Um, 31 against 29 in favor. 29 υπέρ 29 κατά. Άρα απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την... Α, όχι. Μπορείτε να δείξετε το αποτέλεσμα πάλι παρακαλώ. Τροπολογία 229 υπέρ. Κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Both is closed. Τέλος Απορρίπτεται. Βλέπετε τα αποτελέσματα, ωραία. Τροπολογία 231 και 230 και όχι. 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.30 είναι ταυτόσημη πάω στη 2.32 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Στη 232 ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 19 ψηφίζουμε Vote is closed is adopted. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 20. Both is closed. Τέλος της Εγκρίνετε. Εγκρίνεται. «239». Τροπολογία 239. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Συγγνώμη, αλλά είναι πολύ ε, ε, σφιχτές οι ψηφοφορίες, οπότε πρέπει να ελέγχουμε. Ψηφίστε παρακαλώ, τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική σε ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται C2 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη C2 Vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβιβαστική C υπέρ Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την C. Συμβιβαστική C. Ψηφίζουμε και ηλεκτρονικά για τη συμβιβαστική C. Τέλος ψηφοφορίας. Έκρινεται Με μεγάλη πλειοψηφία, επιτέλους. Λοιπόν, συμβιβαστική D. Με προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπάρχει αντίρρηση. Στην προφορική. Τέσσερα χέρια χρειάζονταν για την αντίρρηση. Ωραία, οπότε δεν, δεν θα γίνει αυτή η προφορική. Ψηφίζουμε λοιπόν στην συμβιβαστική ε λέει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Όχι, για την D με συγχωρείτε. Ε, συμβιβαστική D ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ένας ακόμα πρέπει να ψηφίσει. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται... Uh, D1. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβιβαστική D1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική D2. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οπότε τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την 265. Σωστά. Τροπολογία 265. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 265. Still want to vote? Vote is closed. Τέλος της πληροφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 266. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για τη 266. Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Is rejected. Yes. Now we vote to 267. 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 268 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 268 Vote. Vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. So, sorry, we reopen the... Ναι, συγγνώμη, να ξαναψηφίσουμε λοιπόν γιατί... 2.68, ποιοι είναι υπέρ. Όχι, συγγνώμη, ήμασταν στον ηλεκτρονικό έλεγχο. 268 vote is open. Still two people to vote. Δύο ακόμα δεν ψηφίσατε. Ψηφίστε παρακαλώ. Γιατί 268. Okay, vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 268 εγκρίνεται. 269. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Vote is Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2,70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Συμφωνήσαμε ότι υπάρχει μια σειρά. Ακολουθήστε τον Πρόεδρο. Ε1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε2 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την ε2. Still want to vote? E2. Okay, vote is... Ωραία, πέρασε ψηφοφορίας απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την Ή, την Ε, υπέρ κατά αποχές, έλεγχος για την Ε, ε συμβαστική Ε. Vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Του, άντε πάλι μία-μία. Of Fulvio... 2.75. Φούλβιο Μαρτουτσέλο. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 278 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 278 Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 279 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για τη 279. Α, συγγνώμη, πρέπει να επαναλάβουμε την, την ψηφοφορία γιατί υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Α, και εγώ, ναι, μάλιστα. Δύο συνάδελφοι. Γιατί πρέπει να ξαναψηφίσετε, γιατί έκανε λάθος και ακύρωσε το μηχάνημα. Δύο δεν θέλετε να ψηφίσετε. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 2.79. Αν εγκριθεί, πάμε στη 2.76. Ποιοι είναι υπέρ της 2.76. Κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε πάμε στην 274 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη 274. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για τη 274. Έχουμε δημιουργικού συνδυασμού στην ψηφοφορία μας. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται αυτή. Λοιπόν, περνάμε στην 282. Υπέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 284. Υπέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 283. Υπέρα. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 286. Υπέρα. Κατά. Αποχές Έλεγχος για τη 286. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ε, τώρα πρέπει να πάμε στη 288. 288. Οι 289 και 290 καταπέπτουν. Αυτό είναι παράξενο γιατί δεν αναφέρονται σε αυτές που καταπίπτουν. Μάλλον δεν υπάρχει κάποιο λάθος. Θα τις ψηφίσουμε. 2, 8, 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2,90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2,88 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος για τη 288. Ψηφίζουμε. Α, ήσασταν πολύ γρήγορο. Πολύ ωραία, εγκρίνεται. Πάμε στη 292. 371. Ψηφίζουμε για τη 371. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 372. Unblock με την 687. Α, έχουν καταπέσει. Οπότε πάμε στην 685. Ωραία. 685. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 688. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ο Μπούρκαρ το καταψηφίζει τον εαυτό του. Πάμε στο 689 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 686 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 294 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 295 υπέρ κατά υπέρ, υπέρ κατά Αποχές. Έλεγχος για τη 295. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική F1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. F2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την F2. Τέλος της πληροφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική F. Περ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την F. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 304. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 300. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 300. Ψηφίζουμε. Τέλος πληροφορίας απορρίπτεται. 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 331 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 308 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Εγκλέγξουμε το 308. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλο τη closed. Απορρίπτεται. 350 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά ας το ελέγξουμε γιατί δεν είμαι σίγουρος. 350 λοιπόν. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Closed is rejected. 320. 323 ε, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 323. Ένας ακόμα πρέπει να ψηφίσει. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 322 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω τα χέρια σας ξανά λοιπόν 322 ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ πέρας τις οφορίες. απορρίφθηκε 310 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται εκτός αν θέλετε να ελέγξουμε όχι 309 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 309 μπορείτε να ψηφίσετε Πέρα της σοφορίας απορρίφθηκε 311 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 312. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ηλεκτρονικά νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά ελέγχουμε 312. Ψηφίστε. Πέρα της φοφορίας. Απορρίπτεται. 313. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 314 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 316 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 318 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 318. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άλλος ένα πρέπει να ψηφίσει. Εντάξει, πέρα τη οφορίες. Απορρίφθηκε. 319. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 319. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Είναι συμβατή η 317. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 317. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 324 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 335 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. 335 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Άλλος ένας μένει. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 326 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 327. όχι, είναι ίδια. Είναι ίδια. 328 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 300. Όχι, είναι ίδιες. 332. 332 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε για την 332. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τις οφορίες. Απορρίπτεται. 333 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 333. Ψηφίστε. Πέρα τις οφορίες. εγκρίνεται. 336 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. 336 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Α, όχι, κατά πι, τι είπαμε 334, 336 ψηφίζουμε. Πέρας της οφορίας εγκρίθηκε. 337 τώρα. Υπέρ 337. Για άλλες καταπίπτουν. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 338 είναι η ίδια. Πάμε στο εισηγητού, την 27. 27 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 27. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της οφόριας, Απορρίπτεται. 347 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για 347. Ψηφίστε. Πέρας της οφόριας, Εγκρίνεται. 348 υπέρ. Κατά. Αποχές Να ελέγξουμε. Ωραία. 348. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Άλλος ένας. Πέρας της οφορίας. Εγκρίνεται. 351 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε. 351. Ψηφίστε παρακαλώ. Αυτό πέρα της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 352. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 353. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 354 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 355 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. 355. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Α, όχι, όχι, απορρίπτεται. Είδα τώρα καλύτερα ποια ομάδα ψηφίζεται. Απορρίφθηκε. Ωραία. 356. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. 356. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 357. Υπέρ κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. 357. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της οφορίας απορρίφθηκε. Συμβιβαστική F α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. F A. F α. Ψηφίστε παρακαλώ. Συμβιβαστική. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική G1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική G. Κατά δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της οφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική H1. Ήτα 1. τα 1 Κατά. Αποχές Ελέγχουμε για την ΙΤΑ 1, H1. Ψηφίστε παρακαλώ. Άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική H, ήτα, υπέρ, της φοφορίας. απορριφθηκε συμβαστικη h αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική I1. Υπέρ. Α, έχει αποσυρθεί. Αποσύρθηκε. Και οι τρεις τροπολογίες οι προηγούμενες, γι' αυτό είμαστε στην I1, J1 δηλαδή αντίστοιχα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική I. Υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε τη συμβαστική I. Υπέρ, να ψηφίσετε μάλλον ηλεκτρονικά. Πέρα της φοφορία Εγκρίθηκε. Συμβαστική J. Υπέρ, κατά, αποχές ελέγχουμε συμβιβαστική J. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική K1. K1 στη σελίδα 17 στο δικό μου το κατάλογο λέει ο πρόεδρος Γυρίστε μερικές σελίδες. Σελίδα 17, συμβιβαστική K1. K1. Το βρήκατε? Γυρίστε τις σελίδες. Περιμένω, ναι. K1 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική K2 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. K2, K2. Ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Πέρας της απορίθηκε απορρίφθηκε. Συμβαστική K, υπέρ. Κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Συμβαστική K, Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της σοφορίας απορρίφθηκε. Συνεπώς, Α, νόμιζα ότι είδατε το αποτέλεσμα. Ορίστε, παρακαλώ να δούμε το αποτέλεσμα στην οθόνη. Διαβάζουμε. 30 κατά, 29 υπέρ, μία αποχή. Δεν ξέρω γιατί δεν φαίνεται, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αν κοιτάξει κανείς απάνω, θα το δει. Θέλετε να το δείτε. Να. Θέλετε να πάρετε φωτογραφία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Καλώς. Παρακαλώ κύριε Λάμπερτς. Σαν διαδικαστικό. Δεν είναι η πρώτη συμβαστική πρόταση που απορρίφθηκε. Όλες ε, απορρίφθηκαν λίγο πολύ στα διάφορα άρθρα. Και ανησυχώ γιατί θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου ψηφίζοντα τροπολογία-τροπολογία θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο που δεν θα έχει συνοχή. Και δεν μιλάω τώρα υπέρ ή κατά. Απλώς με το αποτέλεσμα. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα μας κάνει να φαινόμαστε γελοί. Είπαν κάποιες ομάδες ότι θέλουν σήμερα να ψηφίσουμε, αλλά αυτή είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που μπορεί να μας οδηγήσει σε αχαρτογράφητα νερά. Πρόεδρος, η προειδοποίηση που μας στέλνετε είναι σοβαρή. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί παρουσιάζοντας τις θέσεις μας. Δεν το βλέπω όμως και βλέπω ήδη να υπάρχει δυσκολία για να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό κείμενο. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Παρακαλώ κυρία Φερέιρα. Εγώ απέφυγα να το πω, μιας και το είπα στην αρχή, αλλά υποστηρίζω το σχόλιο του κ. Λάμπερτς, διότι χάνεται οποιαδήποτε συνοχή, ε, η συνοχή δηλαδή σε ένα τέτοιο συνεκτικότητα, αν θέλετε, σε ένα τέτοιο κείμενο, όπως ψηφίζεται τώρα, θα τίνει προς τα μηδέν. εγώ νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, συμφωνώ μεν. Με όσους λένε ότι δυσχεραίνεται κάπως η κατάσταση διότι απορρίπτονται οι συμβασμοί, σε ορισμένε περιπτώσεις επιστρέφουμε στο αρχικό κείμενο της Κομισιόν, αλλού πάμε σε επιμέρους τροπολογίες που έχουν υποστηριχτεί. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν κάπως καλύτερα σε ό,τι αφορά τους συμβασμούς, εγώ πάντως προτείνω να προχωρήσουμε. Πρόεδρος Γκουαλτιέρη, τα σημειώνω. Ε, συμφωνώ βεβαίως με την ανησυχία του ε, κύριο Λάμπερτς, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Το 488, υπέρ. Κατά. «488» επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Αφού η συμβαστική κάπα έχει εκπέσει και έχουμε τώρα την 488. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 490. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 492. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. 501. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 502 υπέρ κατά αποχές

Ναι, ναι, ναι. Εγκρίνεται λοιπόν συνολικά. Α, ξέχασα τις αποχές λοιπόν. Εγκρίνεται λοιπόν. 503 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. 504 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Αφού είναι όλες ταυτόσιμες, πηγαίνουμε 45 υπέρ. Κατά αποχές. Επαλήθευση. Τέλος. Εγκρίνεται. 511 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 512 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση αρχίζει Απορρίφθηκε 511. Γι' αυτό ψηφίζουμε την 512. Τέλος. Εγκρίνεται. 46 είναι συμβατή. Άρα η 46 ψηφίζεται. Υπέρ, κατά, αποχές. Επαλήθευση. Ακόμα τρεις δεν έχουν ψηφίσει. Τέλος. Εγκρίνεται. 513. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Εγκρίνεται. 514 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 525 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 517 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 522 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Τέλος. Εγκρίνεται. 521. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Τέλος. Απορρίπτεται. 5.19 και 5.20. Υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνονται. 516 υπέρ, κατά αποχές. Επαλήθευση. Εκπίπτει, λέει ο πρόεδρος. Α, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. 518. 518 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 526 υπέρ Α, μαζί με την 527 και 28 και 2.38. Όλες μαζί. Στη λίστα μου βλέπω και 238 λέει ο Α, χωριστά. Ωραία. Α ψηφίσουμε χωριστά. 5, 26, 27, 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Τέλος. Εγκρίνονται. 238. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 529 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 532 υπέρ. Κατά αποχές. Επαλήθευση, λέει ο πρόεδρος. Αρχίζει. Τέλος, εγκρίνεται. Πεντακόσια τριάντα υπέρ. Κατά. Αποχές. 532 ξανά την αρχή. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 538 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Τέλος, εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 48. Πέρας. Εγκρίνεται. 5.39 υπέρ. Κατά. Αποχές. 539 επαλήθευση. Τέλος, Εκκρίνεται. 540 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 541 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5.42 και 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5.45 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται επαλήθευση 545 Εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. 546 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 548 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 549 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 551 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 552 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 553 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Τέλος εγκρίνεται. 5.54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 555 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 556 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την 50, να αρχίσει η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίθηκε. Συμβιβαστική L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική M υπέρ υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Συμβιβαστική M ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της σοφορίας εγκρίθηκε. Συμβιβαστική ένα N υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε τη συμβαστική 1, νη. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της οφορίας, εγκρίθηκε. Τροπολογία 641, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 652 υπέρ, Α, 642 διορθώνει ο πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 643 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την 55. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις οφορίες απορρίφθηκε. 644 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 644. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της Απορρίφθηκε. Πρόεδρε, νομίζω ότι έχει γίνει ένα λάθος τεχνικό για την 55. Μήπως θα μπορούσαμε να ξαναψηφίσουμε. Όχι, λοιπόν, ο Πρόεδρος, ψηφίσαμε ήδη. Έπρεπε να το είχατε πει νωρίτερα, αλλιώ θα χαλάσουμε μια αρχή που έχουμε. 645 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίφθηκε νομίζω, αλλά ελέγχουμε για την 645. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις οφορίες απορρίφθηκε. 646 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την 56. Ψηφίστε παρακαλώ. Άλλος ένας πρέπει να ψηφίσει. Πέρας της οφορίας. Εγκρίνεται. 56. Ήταν αυτή. 647 είναι συμβατή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω. 57. Υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε. 57. Ψηφίστε παρακαλώ. Απορρίφθηκε. 30-30. 648 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 649 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. 58, πιστέψτε με, εγκρίθηκε, αλλά εντάξει, ελέγχουμε. Άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Πενήντα Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε για την 59. Και οι υπόλοιπε είναι μια ομάδα τροπολογιών που είναι ίδιες μεταξύ του. Λοιπόν, ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν. 654 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Πι. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 670. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 671 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 672 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. 672. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 673. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, απορρίφθηκε θέλω να πω, απορρίφθηκε βέβαια. 674 είναι ίδια, έτσι, ωραία. 675 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 676. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 677. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε. 677. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της οφορία απορρίφθηκε. 678 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 601 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 680 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 681 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 682 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 682 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε της φοφορίας απορρίφθηκε. 63 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε 63. Ψηφίστε παρακαλώ. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 684 είναι συμβατή υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 684. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 690. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 691. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 692. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 744 υπέρ, α, μαζί με την 183 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται νομίζω. Εκτός αν θέλετε να ελέγξουμε. Καλά, σε ελέγξουμε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκαν. 746 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. 65 ελέγχουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 747 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε για την 66. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίθηκε. 749 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 750 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε 750, ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Απορρίφθηκε. 68 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε για την 68. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της οφορίας, εγκρίθηκε. 751 υπέρ. Α, συγγνώμη. Καταπίπτουν. 753 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την 69. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Η διερμηνία σταματάει για τη συνεδρίαση αυτή. Abstentions. Again, check. 70. Vote is open. Three people to vote. Vote is closed.